Ακριβώ για να προσθεθούν αυτοί και θα πρέπει να δούμε την συναπόφαση μέσω των εργαζομένων πάντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τίνει προ ένα πιο κοινωνικό χώρο και μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει αλλά όχι πλήρω ε, και στα πλαίσια της του 2020 και μαζί να συμμετάσχουν εταιρείε. Θα πρέπει να οι προσπάθειε ώστε τα εμπόδια να καταπέσουν σε εταιρική αγορά αυτά που εμποδίζουν την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σεβόμενοι το δίκαιο των εργαζομένων που δεν θα πρέπει να είναι τα θύματα της μεταφοράς αυτής των εταιριών αλλά ε, να κερδίσουν και αυτοί όπως και οι εταιρείε ε, και να είναι κάτι το πιο ανταγωνιστικό, πιο παραγωγικό ε, και οι εταιρείε θα πρέπει να προσφέρουν θετικά στοιχεία όπως και στην προηγούμενη χώρα που είχαν κατασταθεί ακόμα και καλύτερα και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι κεφαλικές εταιρείε εταιρείε, οι πιο αδύναμε δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τι σημερινέ υποχρεώσει και που παρεμποδίζουν την καλή του απόδοση. Καταλήγοντα ε, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια μελέτη εφικτού και επιπτώσεων σύμφωνα με το σχετικό τη συνθήκη και μετά από την δημοσίευση τη επιτροπή του 2007 ε, σεβόμενοι τα δικαιώματα των εργαζομένων ελπίζουμε όσο πιο σύντομα να καταλήξουμε σε μια ε, καλή ε, κατάληξη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Ρενιέρ και μετά η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά την παρέμβαση του εισηγητή και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια επικοδομητική λύση εδώ στην Επιτροπή μας ακολουθώντας τις γενικές γραμμές που μας έδωσε ο εισηγητής. Νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξεπεράσουμε τις Αντιφάσει που υπάρχουν μεταξύ των νομοθετικών συστημάτων των κρατών μελών. Πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνεται σε περίπτωση της μετακίνησης της ε, μεταφοράς της μεταφοράς της έδρας της μιας Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα βαθμό εμπιστοσύνης και βεβαίω να υπάρχει και το δικαίωμα συμμετοχή ε, και κάλυψη των εργαζομένων. Νομίζω ότι η κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει ο συνάδελφο Μπουλάν είναι ορθή. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει αξιολόγηση αντικτύπου Και βεβαίω και απόφαση για το ποια νομοθεσία θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τη διασυνοριακή μεταφορά τη έδρα αλλά και τη φορολογική έδρα. Νομίζω ότι οι παρατηρήσει του εισηγητή ήταν όλε ενδιαφέρουσε. Απλώ να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία είναι ένα εγχείρημα που κατά κάποιο τρόπο πάγωσε Πιστεύω λοιπόν ότι δεν έχει απαντηθεί επαρκώς το ζήτημα της διασυνοριακής ε, μετακίνησης. Πρέπει το ζήτημα αυτό να αποσαφινιστεί, διότι ακόμη και το θέμα της μεταφοράς έδρας θα... δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Το να χρησιμοποιήσουμε τώρα τα όρια ε, της οδηγίας για τις συγχωνεύσεις, όπως πρότεινε ο εισηγητής, μου φαίνεται κάπως περιοριστικό. Με διάφορες ε, διαπραγματεύσεις καταφέραμε να πετύχουμε ικανοποιητικέ λύσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν προτιμότερο να ακολουθήσουμε αυτές τις ε, κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, για τις δικές σας εισηγήσεις βρίσκονται ότι περισσότερες ήταν αρκετά εύστοχες και θα τις ε, σκεφτούμε με προσοχή. Κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του για την ε, έκθεση αυτή και για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, όπου ε, εργάζομαι ως τακτικό μέλος. Ευχαριστώ τον κύριο Βουλάν για την ε, θετική του προσέγγιση με ισόρροπη αξιολόγηση των δικαιωμάτων εργοδοτών και εργαζομένων σε περίπτωση που μια εταιρεία θελήσει να μεταφέρει την έδρα της. Επίσης, επιμένει στο ότι πρέπει οι εταιρείε να έχουν ελεύθερο δικαίωμα ε, εγκατάσταση τη έδρα του, ανάλογα με την ε, συνθήκη και όλα στι λειτουργίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται εδώ μελέτη αντικτύπου και τον ενθαρρύνω ενεργά να συνεχίσει να δίνει έμφαση σε αυτό το σημείο. Επειδή οι εταιρείε μπορούν να μεταφέρουν την έδρα του μέσω πόλη και δημιουργία νέου νομικού προσωπού σε άλλο κράτο μέλο, είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση έχει αντιμετωπίσει ως τώρα μεγάλους διοικητικούς και γραφειοκρατικούς φραγμούς, περιτά, κέρδη, ε, κόστος και ε, κοινωνικές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το κόστος και να, καθο... να προστατεύσουμε το ε, δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των εταιριών. Επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε στους ε, μετόχους τους πιστωτέ και του εργαζομένους τα δικαιώματά τους σε περίπτωση μεταφορά. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλλω και εγώ όσο μπορώ στο έργο του εισηγητή και θα κάνουμε τις απαραίτητες προτάσεις βάσει του άρθρου 9 της συνθήκη, δηλαδή προώθηση υψηλού επίπεδου απασχόληση, εγγύηση τη απαραίτητη κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο εκπαίδευση και προστασία της ανθρώπινης υγείας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την απόλυτη δεσμευσή μας να προχωρήσουμε με γνώμονα την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Πραγματικά ε, αδειμονώ για την επικοδομητική συνεργασία που θα έχουμε με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους κοιόδης σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και συγχαίρω, συγχαίρω τον κύριο Μπουλάν για το ως τώρα έργο του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι εδώ έχουμε μια ειδική διαδικασία. Δεν είμαι βέβαιο ότι ο καθένα έχει ακόμη αντιληφθεί τον αντίκτυπο. Διότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πρέπει να ετοιμάσει μια γνωμοδότηση νομοθετική. Εξού και διατύπωση της, ε, για σύσταση που εμφανίζεται στο τέλος της ε, γνωμοδότησης. Υπάρχουν άλλες, άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Εάν όχι, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο ή εκπρόσωπο της Επιτροπής. Θέλετε να πείτε κάτι? Φαντάζομαι ότι αν το Κοινοβούλιο ετοιμάζει νομοθετική γνωμοδότηση, το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν έχει κινητοποιηθεί επαρκώ για το θέμα αυτό τώρα. Μάλιστα, η Επιτροπή Σιωπά, ο εισηγητή. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τις κοδίες κοιτρίες για τις παρεμβάσεις τους. Άκουσα τις παρατηρήσεις της κυρίας Ρέκνερ. Σε σχέση με την οδηγία. Όχι αναγκαστικά για τις συγχωνεύσεις, αλλά αυτή που αφορά τους μετόχους και την αξία των μετοχών. Όπως είχα πει προηγουμένως, είμαι πρόθυμος να συζητήσω όλες τις ιδέες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. για το θέμα αυτό. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών καλύπτει και τις διακοπές. 17 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Λίγη προθεσμία. Θα συζητηθούν στις 8 Σεπτεμβρίου. Και στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε, ενώ η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα ψηφίσει στις 11 του μήνα και η Ολομέλεια θα εξετάσει το θέμα το Νοέμβριο, στην πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Κλείνω με το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Για τις ψηφοφορίες, εάν δεν σας πειράζει να περιμένουμε λιγάκι, διότι οι συνάδελφοι έρχονται βάσει του προγράμματος. Την ώρα που προβλέπετε για τις ψηφοφορίες, πράγμα λογικό. Ας επωφεληθούμε λοιπόν αυτό το, αυτό τα λεπτά χαλάρωσης για να πληροφορήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής και επειδή το συζητήσαμε και στη συνάντηση των συντονιστών στα πλαίσια της προετοιμασίας του κοινωνικού G20 που θα οργανωθεί στο τέλος Σεπτέμβρη. Να σας πληροφορήσω λοιπόν ότι αναλάβαμε την πρωτοβουλία να δεχτούμε την πρόσκληση του κυρίου Σωμαδιά, του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Αυτό είναι μια ιστορική στιγμή γιατί είναι η πρώτη φορά που θα λάβει το λόγο στα καθήκοντά του αυτά στην Ολομέλεια του σώματός μας. Βέβαια ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του ε, σώματος θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες ειδικέ διευθυντήσεις για να οργανωθεί η παρέμβαση του κυρίου Σωμάδια. Θα πρέπει να διακοπεί δηλαδή η Ολομέλεια στο Στρασβούργο την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία μιλάμε για τις 14 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, διότι ο κανόνας προβλέπει ότι σε μία επίσημη σύνοδο μπορούν να παρέμβουν μόνο αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ή ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ. Έτσι λοιπόν θα επιτρέψουμε στον κύριο Σωμάδια να, παραστεί στην, να παρέμβει μάλλον στην Ολομέλεια με διακοπή της Ολομέλειας που εκείνη τη στιγμή θα μετατραπεί σε διάσκεψη των Προέδρων όπου θα είναι προκεκλημένα και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Έτσι θα μπορέσει ο κύριο Ομάδια να λάβει το λόγο στην Ολομέλεια και ο καθένα να συζητήσει μαζί του κάτι που νομίζω είναι και ο στόχο όλων μα. Εάν δεν τα οργανώναμε έτσι τα πράγματα, γιατί βέβαια μπορεί να έχουμε και πρόοπτα στις 14 Σεπτεμβρίου, σε αυτή την περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα θα διοργανώσουμε, θα προβλέψουμε μάλλον την υλοποίηση των προτάσεων μεταρρύθμισης που επεξεργάστηκε ο συνάδελφος Βόποντα, Δηλαδή, τον κανόνα που προβλέπει κοινή συνάντηση στο ημικύκλιο με την ε, Επιτροπή. Τη δική μας Επιτροπή και όλων των Επιτροπών ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2011, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας θα βρίσκεται ε, εντός των τυχών και θα μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση μαζί του. Ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω όχι μόνο για να γεμίσω το πεντάλεπτο, αλλά για να κινητοποιηθείτε. Γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική αυτή και για τα θέματα της Επιτροπής μας. Είναι 9 και 26. Προτείνω λοιπόν να περιμένουμε ακόμη 3 έως 4 λεπτά, ώστε να έρθουν οι συνάδελφοι. Εάν έχετε σημεία να θέσετε ποτά διάφορα, μην διστάσετε. Τώρα είναι η στιγμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω, μάλλον βλέπω ότι σχεδόν όλοι έφτασαν. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε. Και στο σημείο 10 ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Χίρς που έχει να κάνει με τον αγώνα κατά της εγκατάλειψης σχολείου. Παράγραφος 1 Συμβαστική λύση α υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική β μετά από την παραγραφό 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με την παραγραφό 1 η 9 της κυρίας Μωρινσαρτιέ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την 1 έχουμε την γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παρφος 2 τροπολογία 13 κύριε Ζαρόκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 2. 16. Thomas Mann, υπέρ. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. 15 Ρενιέ και Στάινρακ. Υπέρ της 15. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 16. Thomas Mann, υπέρ. Κατά. Αποχές κανονικά εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. και αν ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται 17, Τόμας Μαν, υπέρ. Κατά, αποχές, το ίδιο. Εγκρίνεται πράφος 2, τροπολογία Δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Τροπολογία 19, μονασάρτιε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «27» μπορεί να συνδυαστεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 Τόμας Μάνι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 26 μπουλάων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραγωγή 3, τροπολογία 28 της κυρίας Παπαδοπούλου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 29, κυρίας Παπαδοπούλου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται προστριά συμβαστική υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ήταν η ε, η συμβαστική. Παραφος 4, τροπολογία 33, υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 35 της κυρίας Παπαδοπούλου, υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται η 36 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 4 έχουμε την 39 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 5, τροπολογία 43 της κυρίας Μπισότο, η κατά εισηγείται, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η σίγμα τάφ, πέντε ομάδες, την υποστηρίζουν, την συμβαστική σίγμα τάφ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την 5 έχουμε την ε, 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 56 μπουλάν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 57 πλάμ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 58 πλάμ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 59 πλάμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 Helmer. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την 5 τροπολογία 62 του κυρίου Πουπάκη και μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μάλλον παράγραφος 6 τροπολογία 64 της κυρία Μπιζότο προτείνει διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 Χέλμερ υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, απορρίπτεται, εντάξει, εντάξει, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Ίσως ήθελα να ικανοποιήσω τον κύριο Χέλμερ. Λοιπόν, η επόμενη, η ζη λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν πολλές παρακάτω και μετά την 6 έχουμε την τροπολογία την 80 πια του κυρίου Γκουτιέρες Πριέτα και Αλεχάνδρου Θέρκας. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 6, 81, Μπουλάν, αυτή καταπίπτη όπως και η 82 καταπίπτει, 83 της κυρίας Τσίμερ, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 84 Τζίμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 Τζίμερ υπέρ κατά αποχές ε, κανονικά απορρίπτεται να το δούμε όμως ψηφίζουμε και αν ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορία. 28 υπέρ 19 κατά δεν άλλαξε τίποτα, εγκρίνεται. 85 σήμερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 τουρμεν, τουρούνεν, συγγνώμη. Υπέρ Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Επαναλαμβάνω, 84 εγκρίνεται και 85 εγκρίνεται. Την 86 ψηφίζουμε. Υπέρ της 86. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για την 86. Να ελέγξουμε την 86. Ψηφίζουμε. Και αν ψήφισαν όλοι. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 87 τούριν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 τουρούν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 χείρ, υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Παράγραφος 7 η 90 Τσίμερ υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 μπουλάω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 όχι όχι καταπίπτει 94 ψηφίζουμε την 95 πάξας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 του Ρούνεν ναι, συμβατή, αλλά λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 7 έχουμε την 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 καταπίπτει 98 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 μπιζότο υπέρ κατά αποχές για να δούμε την 101 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 101 και αν ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες 24-21 εγκρίνεται 102 τούρνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 του κύριου Πουπάκη και Μπαλντασάρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 Πουπάκη Μπαλντασάρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 του κύριου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 8 107 χείρς του Ρούνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νέα, συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 καταπίπτει Πατρακτό έχουμε την 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραφορσοκτό 8 η 114 καταπίπτει αυτή ψηφίζουμε την 115 Γκουτιέρες και Σέρκας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 9 όχι όχι να ελέγξουμε μάλλον λάθος θα έκανα λοιπόν για να δούμε την 115 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Πέρας της ψηφοφορίας. 21-19. Εγκρίνεται. Μία αποχή. 116 μπιζότο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική η H το λατινικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πράγμα 9. 124 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελευταία 125 του Ρούνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά για την γνωμοδότηση της κυρίας Χίρς. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ε, Ένας από το ΕΛΚ όμως να μην ψηφίσει. Εντάξει. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρα τη ψηφοφορία. 46 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρτήρια στην κυρία Χίρση. Et nous en venons au point 11, au vote. Σημείο 11. Pour la lettre, euh, pour monsieur. Λοιπόν, Έχουμε την επιστολή για τον κύριο Δημοσίου Πρόεδρο τη Επιτροπή για την κινητοποίηση του ε, ε Ταμείου Προσωπική Παγκοσμιοποίηση για την Αυστρία. Δύο επιστολές για την Αυστρία. Έχουμε τα σημεία 11 και 12 δηλαδή στην ε, ψηφοφορία μας και προτείνω να τα ψηφίσουμε και τα δύο μαζί. Καθώ είπε κοινοτοποίηση τεχνική βοήθεια για το 2011. Διαφωνεί κανένα να ψηφίσουμε από κοινού τις τρει αυτέ επιστολέ. Όχι, ωραία. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνονται. Και περνάμε τώρα στο σημείο 13 της τη διάταξη. Ε, πρόταση έκθεση του κ. Λούτβικσον για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Παράγραφ 11. Παράγραφος 11. Η τροπολογία 14 απεσύρθη. Συμβαστική γάμα λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. παράγραφ 1. Μετά την παράγραφο 1. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Για κατατμήματα ψηφοφορία. Όλο το κείμενο χωρίς αυτό των κοινωνικών πολιτικών που σκούν τα κράτη-μέλη. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι ενεκρίθη για να ελέγξουμε όμως. Άρχεται η συμφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 22 υπέρ, 21 κατά, 5 εποχές. Ναι, πραγματικά χρειαζόταν πάντως επαλήθευση. Μετά, τροπολογία 20 του κυρίου ε, Μπουλόν και Μόβεμ Σαχτιέ με μια προφορική τροπολογία που την έχετε πάρει γραπτά. Διαφωνικά με την προφορική τροπολογία. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν την 20 τροποποιημένη υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν, συμβαστική τροπολογία ε υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 22, κορνελίσεν υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Φιγκερέτα Λοϊαρίκ. Με μια προφοβική τροπολογία που συμφωνείτε όλοι με αυτή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, λέει κάποιος από την αίθουσα. Ωραία, να ελέγξουμε για την 23. Tout le monde a pu voter Ψηφίσατε όλοι. Πέρας πληροφορίας. 26 υπέρ, 23 κατά. Είναι κρίθη. Παλιά 24 των ιδίων. Με κατευθύνματα ψηφοφορία. Το σύνολο κειμένου χωρί αυτό που λέει which the τα of the κλπ. κλπ. Υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε καλύτερα. Ψήφισαν όλοι πέρα στι ψηφοφορία. 20 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται, άρα το δεύτερο τμήμα δεν έχει κανένα νόημα. Τροπολογία. 25 για την παράγραφο 2. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασική, δε. Υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 ψυχήτρια. Α, όχι. Η 27 επεσήρθη. Συμβαστική κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Λούτριξον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 του Α, όχι, έχει καταπέσει. Συγγνώμη. Ε, συμβαστική F, σιγματά. Υπέρ. Κατά εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Λιερίκ Φιγερέτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την 3, τροπολογία 40, με κατατμήματα ψηφοφορία. Το σύνολο κειμένου χωρίς το τμήμα αυτό που αναφέρεται υπέρ, κατά, εποχές. Να ελέγξουμε καλύτερα. Τη 40, το πρώτο τμήμα τη 40. Tout le monde a Ψήφισαν όλοι οι πέρα ψηφοφορία. 26 υπέρ, 23 κατά. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, Απαρρίπτεται. Για την παράγραφο 5, εισαγωγικό τμήμα, έχουμε μια συνδραστική τροπολογία άσου. Και εδώ θα καλτώ τη θέση μου ως Πρόεδρο και θα προτείνω μια προφορική τροπολογία, γιατί είπαμε χθε ότι η συμβαστική λύση που αποφάσισαν οι διάφορες ομάδες συμπεριλαμβάνουν τους κοινωνικούς εταίρειους, τον επιχειρησιακό τομέα και τις μη κυβερνικέ οργανώσεις. Και είχα πει χθε ότι αυτό είναι μια επανάληψη. Λόγω των κανόνων στο σώμα δεν μπορούμε να κάνουμε κατά τμήματα ε, ψηφοφορία για να φέρουμε τον όρο business sector. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια προφορική τροπολογία. Αν αφήσουμε τα πράγματα έτσι, έχουμε δύο φορές εκπροσώπηση των ε, εργοδοτών. Και όταν λέμε κοινωνική εταίρη και όταν λέμε στο μέσα. Εάν θέλουμε λοιπόν να το βγάλουμε ή όλες οι ομάδες συμφωνήσουν μεταξύ τους να αφαιρέσουμε αυτό το Business Center ή θα προσθέσουμε τα συνδικάτα. είναι πιο ευρύ το business center, business sector, συγγνώμη, από ότι οι κοινωνικοί εταίροι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε δύο φορές τέτοια πράγματα. Να επαναλάβουμε και τα συνδικάτα. Κύριε Κλάκ. Όχι, ο κύριο Έλμερ. Κύριε Πρόεδρε. Ε, λυπούμε, ίσως κάτι δεν κατάλαβα σωστό. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα, εισαγάγετε μια προφορική τροπολογία. Εγώ είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας, αλλά δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, θα χάσω έτσι και δεν θα, δεν θα επιμείνω. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα δεχτώ αυτή την τροπολογία ως έχει. Ε, συμβαστική τροπολογία, ας, ήταν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 43 είναι κλωσική, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Παράγραφα 5 Β. Συμβαστική Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα, καταπίπτει το δεύτερο. Τροπολογία 49. Κοφεράτη έγκελ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50, μπιζότο, υπέρ, κατά, Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 μπέκερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 με προφορική τροπολογία του εισηγητή που δεν έχει απορριφθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν το 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 κορνελίσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 το Λιουαΐκ κατά τμήμα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Το πρώτο τμήμα 60. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 26 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 61 μπουλόν καταπίπτει όπως και 62. 63 του ίδιου υπέρ, κατά αποχές. Εν... Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι πέρα τη πληροφορία. 19 υπέρ, 30 κατά. Πραγματικά απορρίπτω, λείπουμε κύριε Μπουλό. Δεν είδα καλά. Τροπολογία 64 με προφορική τροπολογία. Α, όχι, καταπίπτει. 67 αποσύρθη και 69 το ίδιο. Και φτάνουμε στις θεωρήσεις 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 για την αιτιολογική σκέψη β. Με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή δεν διαφέρει κανένας. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη γ. Συμβαστική β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12. Η αρήκτη υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται και 13 των ιδίων υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα ψηφοφορία. 40 υπέρ, 4 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. nous en venons à notre dernier vote. Pardon, Monsieur Baldassar. Για την έκθεση Γκίρλινγκ ω ΕΛΚ ψηφίσαμε υπέρ της τροπολογία 59. Αλλά τελικά δεν θα το κάνουμε αυτό, διότι σε αυτή την περίπτωση θα κατέπτε η συμβαστική λύση F. Ε, όμως, η τροπολογία 59 δεν αντικειτώ το τόσο φανερά στην ε, συμβαστική λύση ΕΦ. Τελικά, έτσι όπως έχει ετοιμαστεί ο κατάλογος πληροφοριών, είναι αντιφατικός και αυτό δεν είναι πολύ λογικό. Τέλος πάντων, την τροπολογία θα την υποβάλουμε και στην ΕΜΚΟ για να παραμένει το περιεχόμενο της 59. Κύριε Βαλτασάρε, σας κατάλαβα σωστά. Είπατε ότι αποσύρετε την υποστήριξη ομάδα σας για την τροπολογία ε, F για να υποστηρίξει την 59. No, Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Η τροπολογία 59 δεν μπορεί να υπερψηφιστεί. Εάν την ε, ψηφίζαμε, δε, μάλλον θα πέρναγε οπότε θα κατέπιπτε η συμβαστική F. Όχι στην 59. Υπάρχει απλώ μια διαφορά στο, στους δημόσιους διαγωνισμούς και στο μέγιστο όριο. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί ετοίμασε έτσι τον κατάλογο ψηφοφοριών η ε, γραμματεία. Ουσιαστικά είναι συμβαστή η 59 με τη συμβαστική F. σω ε, την επόμενη φορά να είστε λίγο πιο προσεκτικοί Τέλο πάντων, εμεί την ιδέα που θέλουμε θα την εκφράσουμε στην τροπολογία που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ήταν απλώ μια διευκρινήση. Ε, θα, ένα δευτερόλεπτο για να εξετάσω ει βάθο το πρόβλημα. Λοιπόν, η τροπολογία 59 της κυρίας Στάινρουκ λέει τονίζει ότι η σημασία ε, ε, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να εξεταστεί ε, πιο έντονα και τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να παίξουν η ε, χαμηλότερο ρόλο στην χρήση. Ο συμβασμός λέει ότι η έλεγχη στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να διευκολύνει τους κανόνες αυτούς και να φροντίσει ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται για τη συμμετοχή στη διαδικασία δημοσίων συμβάτων ώστε να προωθηθεί κοινωνική, περιβαλλοντική και καινοτομική πτυχή τους. Δηλαδή, το να ελισταπιστούν οι διαπατήσεις για τις επιχειρήσεις είναι το ίδιο είναι ισότιμο ότι όταν λέμε θα πρέπει να ενδυναμωθούν γιατί για να είναι συμβατές οι δύο αυτές προτάσεις θα πρέπει ή να τροποποιήσουμε το συμβασμό περιμένετε να δούμε σκέφτομαι μεγαλόφωνα αυτή τη στιγμή Madame 59. Λοιπόν, μήπως μπορούμε να συμφωνήσουμε. Να τροποποιήσουμε τον συμβασμό και να πούμε Μα... Δεν σας έδωσα το λόγο ακόμα. Δεν σας έδωσα το λόγο. Ας κοιτάξουμε πρώτα και μετά θα βρούμε τη λύση. More flexible θα τις πιο ευέλικτες. Αφενός. Είμαι ένα από τους σκιώδεις συζητητέ στην ΕΚΟ και θα να σα πω ότι καταρχήν τα δύο κείμενα είναι πλήρως συμβατά δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να διαθετήσουμε και το ένα και το άλλο εξουσίες. Γιατί στο κάτω-κάτω ήμκο και η Ολομέλεια θα συμφωνήσει μετά. Λοιπόν, ό,τι να προσθέσουμε, και ό,τι βάλουμε σαν σύγχρονα κριτήρια θα πρέπει να βρεθούν και στην ολομέλεια στην ανάγκη. Είμαι σίγουρος ότι τα δύο κείμενα που συζητάμε είναι απόλυτα συμβατά. Madam Πρόεδρε, προσπαθώ να εξοικονομήσω λίγο χρόνο στην συζήτηση γιατί είμαι σίγουρος ότι η συζήτρια δεν θα ήθελε να τροποποιηθεί μια συμβαστική τροπολογία με μια προφορική. Λοιπόν, θα έλεγα, αν δεν διαφωνείτε, να συνεχίσουμε αυτή τη στιγμή και να μην προσπαθήσουμε να αλλάξουμε μια συμβαστική που έχει συμφωνηθεί ήδη. Κύριε το θέμα δεν είναι κατά πόσο θα το τροποποιήσουμε ή όχι. Σε μια συζήτηση υπάρχουν πολλά διακυβέρματα και θα πρέπει να βρούμε την ιδανική λύση. Το πρώτο θέμα είναι κατά πόσο θα τροποποιήσουμε τη συμβαστική τροπολογία. Το δεύτερο είναι κατά πόσο θα θεωρήσουμε ότι αυτέ οι δύο τροπολογίε είναι συμβατέ εν αντιθέσει προ αυτό που έχει αναφέρει εδώ η ε, γραμματεία. Ο κ. Σέγγελ μου είπε ότι θα ήταν καλό να εξετάσουμε τον κατάλογο ψηφοφορία. Αλλά ήθελα να δώσω το λόγο στους τρία άτομα που το ζήτησαν και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Μπαλτασάρ και μετά στην Βεν Ο... Ο συνάδελφος της σωστά ανέφερε αυτό που λέγαμε κι εμείς. Δηλαδή για τα μέγιστα όρια. Η ιδέα αυτή που αναφέραμε, όπως την αναφέραμε, ήταν, ε, μπορούσε να περάσει μαζί με την ΕΦ. Όμως η γραμματεία έτσι όπως τα παρουσίασε τελικά γίνονται αντιφατικά τα δύο μεταξύ τους. Λοιπόν, την επόμενη φορά, εάν προσέξουμε, δεν λέω να τροποποιούμε συμβιβαστικές προτάσεις, αλλά να μην βρίσκουμε και συμβιβαστικές μεταξύ τους λύσεις. Τώρα, εφόσον έχει επιστοποιηθεί, έχει περάσει, εντάξει. Αλλά στην ΙΜΚΟ ελπίζουμε ότι η ιδέα μας στις τροπολογίες 59 θα γίνει δεκτή. Steven Hughes. Κύριε κύριος Χιούς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ναι. Ζήτησα στο λόγο γιατί θεωρούσα ότι θα υπήρχε διαφωνία για την προφορική τροπολογία. Μα δεν χρειάζεται. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ρασιοφορές και να προσθέσουμε την 59 στην συμβαστική. Θαυμάσια. Άλλος που θέλει το λόγο παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Θέλετε πάλι το λόγο εκεί πίσω. Ναι. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι και στις διαπραγματεύσεις είπαμε ότι θεωρήσαμε ότι είναι συμβατές αυτές οι δύο τροπολογίες και θέλω να ψηφίσουμε και τις δύο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει αντίφαση και θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τον κύριο για αυτό που είπε. Θαυμάσια. Η μόνη τροποποίηση για το κατάλογο ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σα είναι ότι εκεί που λέγεται ότι η ψηφοφορία για την 59 θα οδηγήσει στο να καταπέσει η συμβαστική, αυτό δεν είναι σωστό. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε και τις δύο. Συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση έκθεσης της κυρία Ζουλή Γκέρλινγκ για τον εξορισμό τη πολιτική δημοσίων συμβάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που κάνουμε για την ε, ΙΜΚΟ. Υπέρ τη ΠΡΟ 1. Κατά αποχέ. Η συμβαστική Α εγκρίνεται. Τροπολογία 3 είναι συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 Στάινρουκ, συμβατή, υπέρ, Bien, alors, euh, la liste de vote n'indique pas clairement. Λοιπόν, κατάλογο ψηφοφορία δεν λέει ξεκάθαρα ποια είναι τα τμήματα που καταπίπτουν. Με την τροπολογία 6 Μπαλτασάρ, θα πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, που είναι συμβατό με τη συμβαστική. Ποιο είναι υπέρ του δεύτερου τμήματο τη τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, Έντρουεκ. επίση συμβατή, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται, ξεκάθαρα. Τροπολογία 4. όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. 7. 7 του Ρούνου, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριβδόται. Τροπολογία 4. Κάσλερ. Να ελέγξουμε για την 7. Ωραία, να ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι πέρα στι ψηφοφορίε. Ένα από το ΕΛΚ πρέπει να φέρει στην κάρτα από το μηχάνημα. Ακόμα. Εντάξει τώρα. 22 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται, ξεκάθαρα. Τέσσερα λοιπόν. Κάστλερ. Πρώτο τμήμα και δεύτερο είναι συμβατά και τα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 4. Υπέρ. Κατά άποχε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Του Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Του Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Του Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 χιούς και άλλων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κάναμε τροπολογία 22 των ιδίων σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 σε δύο τμήματα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 Είπε. κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συγγνώμη, ενεκρίθη ήθελα να πω. 25 Βαλτασάρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 29, Παλτασάρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31, Παλτασάρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4, 39 σε δύο τμήματα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρέπτεται Σύμβαση απολογία ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Amendement 47 est compatible, je le mets aux voix qui est... 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 καταπίπτει. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 Λούτβιξτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά Λοιπόν, τροπολογία 59. Ε, επαναλαμβάνω ότι το ΕΛΚ είναι υπέρ τη 59 τελικά. Je rappelle que le PPE est favorable à cet amendement 59. Si vous voulez, je ε, κοιτάξτε, μπορώ να γίνω φερέφωνο άλλων ομάδων. Ε. ε λοιπόν. 59. Ποιος είναι υπέρ τη 59. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ξεκάθαρα. Συμβαστική F. σύγματα. Που είναι συμβατή με αυτή την 59 που ψηφίσαμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 του Ρήναν υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιος είναι υπέρ της 58 παρακαλώ. Κατά της 58. Αποχές. Απορρίπτεται. Να αλλάξουμε ευχαρίστω στο 58. Le, le Πέρασε ο 21 προς 28. Πραγματικά απεριφθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν. Την 62 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 63 Μπορούμε να το ζητήσουμε υπέρ, κατά, απαχές απορρίπτεται. 64. Με μια προφορική τροπολογία του κύριου Μπουλό. Δεν διαφωνεί κανένας. Ο κύριος Μπουλό έχει το λόγο, παρακαλώ. Υπάρχει ένα σφάλμα για το ΕΡΚ, νομίζω, στο κατάλογο ψηφοφορία. Δεν τροποποιήθηκε. Είμαστε υπέρ. Υπέρ, το ΕΡΚ υπέρ. Είσαστε σίγουρος, λέτε, ότι σα στηρίζει η ομάδα σα. Θαυμάσια. Λοιπόν. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 Χιούς και άλλων με προφορική τροπολογία της κυρίας Τούρουνεν. Υπέρ της 67 κατά αποχές απορρίπτεται 68 χιούς και άλλων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην παράγραφο 7 τροπολογία 69 Βυζότο για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 70 απεσύρθη. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Συμβαστική Ζ του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 απεσύρθη. 75. Ρέγνα. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 76 χιούς και ο Άλλαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμπαράγραφο 8 77 Τουρνή για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 Λουδίσον και άλλων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 Βαλτασάρδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 χέντρα είναι συμβατή ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 80 Έχει καταπέσει. Έχουμε 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 του Ρινέν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 χιούς και άλλων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 χιούς και άλλων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 Χέντελ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 έχει καταπέσει και έχουμε την 88 Handel υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται 89 πουλό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 του ίδιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 απεσύρθη το σύνολο της πρότασης. Le vote est ouvert. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται. Le PPE, il y a... Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 17 κατά και 4 αποχές.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

ναι, να επαναλάβουμε, να δουλέψουμε και πάλι, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά σημεία στην ημερησία διάταξη, έχουμε πολλά σημεία και πάμε στο σημείο 15, μάλλον για το σημείο 15. Ο κύριος Κοφεράτη θα μας πει μερικά πράγματα για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση. Έχει το λόγο ο εισηγητής μας λοιπόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ύφος των τροπολογιών τους, για το περιεχόμενό τους που έδωσαν και νομίζω ότι σχεδόν στο σύνολό τους είναι στο πλαίσιο των όσων έχω σκεφτεί και εγώ και σίγουρα αυτό θα διευκολύνει τις εργασίες μας. Θα είναι αποτελεσματικότερο, θα είναι δε καλύτερο το τελικό συμπέρασμα. Όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, ένα μέρος αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει στη καθήκοντα της Επιτροπής Πολιτικών Ευθυριών και ε, αυτά που είδαμε είναι θέματα που κανονικά πρέπει να απασχολήσουν αυτή την Επιτροπή. Άρα λοιπόν θα γίνει εκεί η προσπάθεια ξέβρεση συμβαστικών λύσεων. Αλλά είναι ιδιαίτερα θετική αυτή η ιδέα, γιατί κατάλαβαν οι συνάδελφοι το πνεύμα της πρότασης. Υπάρχει διάθεση λοιπόν να εργαστούν όλοι για τη βελτίωσή της και για την ενίσχυσή της. Βέβαια υπάρχουν μετά προβλήματα σύνταξης, ε, διατύπωσης κλπ. Αυτά τα θέματα θα τα λύσουμε και θα μας βοηθήσουν με την ε, πολύτιμη συνεισφορά τους οι σκιώδεις συγητές να υποφεληθώ τώρα για να υπογραμμίσω μερικές πτυχές που κατά την άποψή μου είναι σημαντικές. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάρουν την τελική τους μορφή. Το πρώτο τι αφορά τον, τον τομέα εφαρμογής όλων αυτών. Θα πρέπει να το επαναλάβουμε να το επιβεβαιώσουμε και μετά από αυτές τις τροπολογίες. Δηλαδή, ότι χρειάζεται να βρούμε ακριβώς ε, ιδιαίτερα συγκεκριμένα όσο γίνεται καλύτερα τους τομείς εκείνους ε, στους οποίους θα εφαρμοστεί η οδηγία. Είναι ιστορικά παγιωμένοι αυτοί οι τομείς ε, ακριβώ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό αυτοί οι εποχιακοί εργαζόμενοι και από το βορρά στο νότο έχουμε διαφορετικές εποχές. Γι' αυτό λοιπόν λογικό είναι να σκεφτεί κανείς μια κάποια ευληγησία και ευκαμψία που θα πρέπει να διαθέτουν τα κράτη-μέλη αλλά σε συνόηση ιδιαίτερα στενή με, τις, με τους εταίρους, με όλους. Και έτσι να έχουμε μια ιδιαίτερα καθορισμένη τελική μορφή και μετά δούμε και τις ειδικέ πτυχές που θα εμφανιστούν ε, στις διάφορες χώρες και που θα συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και να δούμε ίσως κάτι που θα μπορούσε να προσθεθεί ακόμα. Δεύτερο θέμα, σημαντικό κατά την άποψή μου σε πολλές πτυχές του, είναι το να εξασφαλίσει κανείς σε όλους αυτούς τους εποχιακά εργαζόμενους τις ίδιες συνθήκες, ε, την ίδια σώρος αμοιβή ε, και συνθήκων εργασίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και έτσι από την συλλογικές συμβάσεις να διαπονται οι συμφωνίες αυτές ε, και να δούμε το μέρος αυτού του σχεδίου. Η συλλογική σύμβαση βέβαια έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική μορφή από τη μία στην άλλη την ευρωπαϊκή χώρα. Αποτελεί όμως το κύριο εργαλείο και υποστηρίζεται αρκετές φορές και από τον νόμο για να καθορίσει τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται τα άτομα αυτά. δεν θα πρέπει να έχει δε, τόσο τρομερό πια βάρος. Αυτή είναι η ανησυχία που εκφράστηκε εδώ, ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι θα μπορούσαν να, καταλάβουν χώρο και θέσεις εργασίας που κανονικά θα έπρεπε να απευθύνονται αυτές τις θέσεις εργασίας σε ντόπιου εργαζόμενους. Αυτό ιστορικά δεν έχει συμβεί. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί και στο μέλλον γιατί έχουμε μέσα για την αγορά, για κάτι τέτοιο, χωρίς να γίνουν ε, δεσμευτικά, χωρίς ε, να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά. Θα πρέπει να δούμε προληπτικά τι μπορεί να γίνει βέβαια, βασιζόμενοι στην πείρα που διαθέτουμε και σε όλα αυτά που γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν έλεγα ίσες δυνατότητες συνθήκες είναι και για την εργασία αλλά και στη ζωή τους, ε, την καθημερινή. Εδώ θα πρέπει να δούμε δύο κύρια σημεία. Πρώτα απ' όλα τη σχέση τους ανάμεσα αυτούς τους εργαζόμενους, εργαζόμενες και τη σχέση τους με τον τόπο καταγωγής τους, προελευσής τους, με τις οικογένειές τους και επίσης ε, η που θα μένουν ε, και το πλαίσιο αυτό που είναι κάτι το πολύ σημαντικό σαν συνιστόσα και συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής ε, αυτών των εργαζομένων. Λοιπόν, υλικές συνθήκες, ενιαία κοινωνική προστασία και επίσης να εξευρεθεί μια κατάλληλη λύση όσον αφορά τις πτυχές εκείνες που έχουν να κάνουν με την κατοικία τους και αυτά τα άτομα όσο γίνεται να τα προστατεύσουμε από κερδοσκοπικές ενέργειες που γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών σε πολλές χώρες και στην Ιταλία, τη δικιά μου χώρα και που καθιστούν δύσκολη την ενσωμάτωση αυτών των ε, ατόμων γιατί τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα και όσον αφορά την εργασία τους αλλά και στην καθημερινή ζωή τους σαν πολίτες ε, για το χρονικό και διάστημα που θα παραμείνουν στη χώρα. Τελευταίο είναι κάτι που έχει σχέση σε συνδυασμό με την Επιτροπή Δημοσίων Ευθεριών ε, μαζί με τους συναδέλφους ε, τους και οδησηγητές αλλά σαν επιχείρημα νομίζω ότι ισχύει πάντα, ότι θα πρέπει να έχουμε στενή επαφή με την Επιτροπή ώστε και διαφορετικές αρμοδιότητες και τα όσα δημιουργούνται να μπορούν να εξετάζονται, να επιλύονται χωρίς να δίνουμε όμως διαφορετικές ε, δυνατότητες, διαφορετικούς δρόμους. Και γι' αυτό το να προσπαθεί κανείς να βρει συμβαστικές λύσεις θα ήταν κάτι το θετικό από τη στιγμή που συμφωνούν και οι συνάδελφοι και οι συζητητές να κάνουμε ένα έλεγχο τουλάχιστον ότι αυτές οι βασικές λύσεις έχουν γενικό χαρακτήρα και σε συνδυασμό, σε συνεργασία με συναδελφούς από τη ΛΥΜΠΕ. Και να δούμε ότι Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν, είναι συμβατά με τα υπόλοιπα και μια κάποια συνεργασία και να μην δημιουργούν διαφορές που να δημιουργούν στρεβλώσεις με τη σειρά τους και να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Στη διάθεσή σας είμαι για να ακούσω σχετικές παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να πείτε μαζί με τις τροπολογίες που υποβάλλατε και μετά σύντομα σύντομα θα προσπαθήσουμε να εργαζόμαστε πάνω στις τροπολογίες αυτές καθευτές με τους κοιόδες ηγητές μαζί. Η κυρία Χίρς και μετά η επόμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρους του σκιώδους μας, του κυρίου Χίρς, μερικά σχόλια. Ένα από τα βασικά θέματα του πακέτου για τη μετανάστευση είναι η ποιότητα τη μεταχείριση. Οι δίκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση με του εργαζομένου των χωρών σε ό,τι αφορά τι ε, συνθήκε εργασία του. Είναι άκρα σημασία να είμαστε συνεπεί εδώ με του κανόνε που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του δικού τη εποχικού εργαζομένου. Οπότε αυτά θα πρέπει να ισχύουν και για του τρίτου, ε, για του πικού τρίτων χωρών που έρχονται για εποχική εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ε, μόνο έτσι, να, μόνο με αυτόν τον τρόπο μάλλον, θα εξασφαλίσουμε προστιθέμενη αξία στην ε, πρότασή μα. Θα αποφύγουμε κάθε διακρατική μεταχείριση και τη δημιουργία πολλών κατηγοριών εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποχικοί εργαζόμενοι που έρχονται εκτό Ένωση θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όσου έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Η ποιότητα τη εργασία θα πρέπει να αφορά τι εργατικέ συνθήκε, ε, του όρου ε, τη πρόσληψη, τα δικαιώματα της κοινωνικής πρόνοιας, συνταξιοδότησης και περίθαλψης εφόσον φύγουν από τη χώρα υποδοχής τους. Η ίση μεταχείριση είναι καθοριστικό σημείο για να μπορέσει η πρόταση να εγκριθεί μεταξύ των υπόλοιπων ζητημάτων που φύγονται στις τροπολογίες και όπου θα πρέπει να αναζητηθεί συμφωνία είναι ο ορισμός της εποχικής εργασίας καθώς είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να μπορούν να προσθέσουν τομείς μετά από συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους η διάρκεια της παραμονής, διότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τα δικαιώματα που προβλέπονται εδώ για τους εποχικούς εργαζομένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στους εποχικούς εργαζομένους να έχουν ε, το απαραίτητο κατάλημα, ε, φροντίζοντας τα κρατημέλη ή εργοδότες να σέβονται τα όσα προβλέπονται από τους κανόνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή ότι η δημογραφική πρόκληση και οι διαφορετικές ανάγκες της εποχικής εργασίας απαιτούν τη χάραξη μιας εξαιρετικής πολιτικής μετανάστευσης μιας πολιτικής μετανάστευσης εποχικής εργασίας που να επιτρέπει να καλύψουμε τα κενά στο εργατικό μας δυναμικό και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό με τους συναδέλφους ετοιμάσαμε κάποιες τροπολογίες για αυτό το σχέδιο οδηγίας. Κατά την άποψή μας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να καθορίσουν το είδος τις κατηγορίες εργασίας που θα επίπτουν εντός του εποχικού αυτού τομέα. Η εποχική εργασία επηρεάζει δημογραφικά και οικονομικά τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τους επαγγελματικούς τομείς που θα αφορά το σύνολο κανόνων για την εποχική εργασία. Βεβαίως συμφωνώ ότι το κατάλημα και οι κανόνες του είναι σημαντικό στοιχείο της πρότασης, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα παραμένουν όλα αυτά κενό γράμμα, διότι τα πρότυπα διαβίωση θα ερμηνευθούν και θα υλοποιηθούν κατά διαφορετικό τρόπο από τα διαφορετικά τη κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει οι κανόνε που θα προβλέψουμε για το κατάλημα να είναι υπερβολικοί σε σχέση με τα που προβλέπονται για τι αποδοχέ των εργαζομένων, για να μην καταλήξουν και περί τι. Το αν ε, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές ή χαμηλές, αυτά είναι στοιχεία που θα πρέπει να αποφασιστούν κατά περίπτωση. Επίση, η κοινωνική προστασία είναι κάτι που θα πρέπει να το ανελάβουν ω αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Να εφαρμοστεί δηλαδή η αρχή τη επικουρικότητα. Επιπλέον, ε, ο εποχικό χαρακτήρα τη εργασία, η σύντομη διάρκεια παραμονή στην επικράτεια ενό κράτου μέλου δεν θα πρέπει να είναι ε, αφορμή για να προβλέπονται για τους εποχικούς εργαζομένους τρίτων χώρων, ώστε να υπάρχει ίδια κοινωνική ασφάλιση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Όπω λέμε λοιπόν και στο σημείο 14 με την τροπολογία μας θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προβλέπουν τις κοινωνικές παροχές που θέλουν να προσφέρουν στους εποχικού εργαζομένους. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για άριστη αφετηρία. Μπορούμε πραγματικά να εργαστούμε πάνω σε αυτά. Εμείς οι πράσινοι υποβάλαμε πολλές και διάφορες τροπολογίες. Όχι επειδή διαφωνούμε, αλλά επειδή θέλαμε να ασχοληθούμε και με λεπτομέρειες για μερικά από αυτά τα σημεία. Χρειάζεται ξεκινώντας να αναγνωρίσουμε ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι στην Ευρώπη ζουν, εργάζονται με συνθήκες τις οποίες μπορεί να ασκηθεί κριτική. Τους εκμεταλλεύονται πολλές φορές και αρκετοί εργαζόμενοι άλλωστε βρίσκονται εδώ παράνομα αλλά είναι άτομα εργαζόμενοι που τους χρειαζόμαστε και αν θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά εργασίας, πρέπει με τον άνα ή τον άλλο τρόπο να ισχύσει μια νομοθεσία στην Ευρώπη. Και αυτό που προτείνει και η Επιτροπή. Συμφωνούμε, αλλά η πρόταση αυτή χρειάζεται να βελτιωθεί, να αποτελέσει τη πραγματικότητα για τα άτομα αυτά που ζουν κάτω από άσχημες συνθήκες ε, να τους αντιμετωπίζει κανείς εξίσου με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους να μην έχουμε μια πρώτη ομάδα και μια β' ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί το κείμενο της Επιτροπής, η σύνταξή του, οι προτάσεις του και νομίζω ότι ο εισηγητής ήδη επετέλεσε πρόοδο και εμείς θα βοηθήσουμε με τις τροπολογίες μας. Για να ασχοληθούμε τώρα με μερικά συγκεκριμένα σημεία που κατά την άποψή μου είναι ουσιαστικά για την όλη συζήτηση. Να δούμε ποιος μπορεί να θελήσει να ζητήσει μια εποχική εργασία. Πρώτα απ' όλα, προερχόμενοι από τρίτες χώρες που είναι σε ένα κράτος μέλος ε, την άλλη στιγμή ακριβώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να είναι άνεργος και θα πρέπει να το επιτρεπεί να βρει μια εποχιακή εργασία. Δούμε δε σε ποιους τομείς μπορεί να το κάνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι η εποχιακή εργασία έχει να κάνει κυρίως με τον τουρισμό και τη γεωργία για να δούμε πραγματικά θα πρέπει να αποκαλείται εποχιακή εργασία. Τέλος πάντων, συμφωνώ πάντως με τον εισηγητή. Εμείς επιθυμούμε την οδογία αυτή να την περιορίσουμε σε κάποιες τομείς, αλλά χρειάζεται και για κάποια ευληγησία και ευκαμψία για τα κράτη-μέλη. Αλλά εμεί οι πράσινοι δεν ξέρουμε ακριβώ το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι κοινωνικοί εταίροι στην ε, πρόταση του κύριου Κομφεράτη προτείνεται να υπάρξει μια διεύρυνση και σε άλλους τομείς ε, εκτός από τη γεωργία και τον τουρισμό και προτείνουμε να μην γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Δεν είμαι σίγουρη ότι αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση. Οι κοινωνικοί εταίροι επηρεάζουν ε, την κατάσταση. Μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν μαζί τους. Και ακόμα κάτι το σημαντικό. Την ορισμό της συλλογικής σύμβασης. Η πρόταση της Επιτροπής, ε, ίσως ο ορισμός δεν είναι σωστός, ίσως είναι και επικίνδυνος. Αυτό που επιθυμούμε είναι περισσότερη λεπτομέρεια και διευκρινήσεις της τροπολογίες. Για να δούμε. Εξέβρεση κατοικίας, η ποιότητά του πρώτα απ' όλα και πολλές φορές ε, είδα πως έχει κατάσταση στη Δανία. Διαπίστωσα ότι οι ξένοι εργάζονται κατά από δυσμενείς συνθήκες, ε, σε υπόγεια, είναι στιβαγμένοι δε σε καθαρτά διαμερίσματα και γι' αυτό χρειάζεται να επέμπουμε σε αυτό και να εξασφαλίσουμε την ποιότητα. Και ακόμη να δούμε πώς πληρώνονται αυτοί οι εργαζόμενοι και τι ποσοστό πηγαίνει στην ε, στο κατάλημά τους. Ε, και πολλοί λένε ότι α, αυτοί είναι από άλλη χώρα, δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει ενίκιο. Τέλος πάντων, τους αφαιρούν διάφορα ποσά από την αμοιβή τους. Ο εργοδότης όμως τελικά είναι κερδισμένος κατοικία στο κατάλημά τους, τα δικαιώματά τους, οι συνθήκες εργασίας τους που πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εμείς υποβάλλουμε προτάσεις επίσης όσον αφορά τις κυρώσεις, τους ελέγχους, γιατί ό,τι θέλετε μπορούμε να υιοθετήσουμε, αλλά αν δεν υπάρξει η κατάλληλη εφαρμογή, τότε δεν θα έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Να δούμε και τους υπεργολάβους. Αυτό να το εξετάζουμε όπως πρέπει πάνω χάρη στον τομέα των υπηρεσιών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Και για να καταλήξουμε, να σας πω ότι υπάρχουν τρεις σημαντικές αρχές. συ αμοιβή αντιμετώπιση. Επίσης, ε, ο περιορισμός των τομέων απασχόλησης και ιδιαίτερα, ιδιαίτερος έλεγχος ε, για την σωστή εφαρμογή αυτών των οδηγιών και έτσι οι λόγω εργαζόμενοι θα μπορούν να έχουν δικαιώματα στην αγορά εργασία μας, εργασίας μας. Κύριε Όμεν Ρόιτεν και κυρία Πρόεδρε όταν ακούω την κυρία Τούρνεν αναρωτιέμαι μήπως η, η Δανία θα εγκρίνει έστω και ένα ελάχιστο ποσοστό των όσων προτείνουμε. Εδώ, στα πλαίσια αυτά, χρειάζεται να επαγρυπνούμε ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έρχονται και εργάζονται σε ορισμένους τομείς στα πλαίσια της εποχιακής εργασίας εάν τους εκμεταλλεύονται ή όχι. Γι' αυτό πρόκειται. Η πρόταση της Επιτροπής τι μας λέει. Στα πλαίσια του συντονισμού από κοινωνικές πλευρές μαζί με τα κοινωνικά επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται να δούμε εάν, ε, τι, ας πούμε, αν ε, μένουν ε, για έξι μήνες σε άλλη χώρα, τι γίνεται με τις κοινωνικές παροχές, μήπως αυτές μπορούν να πληρώνονται στη χώρα προέλευσής τους. Καταλαβαίνω βέβαια και το διοικητικό βάρος, των όγκο εργασίας, για κάτι παρόμοιο αλλά δεν θα κάνουμε τελικά τίποτα. Η κυρία Τουρούνεν ε, προσπαθεί κάτι να πετύχει βέβαια και να δούμε ο εισηγητής ο οποίος υποβάλλει σωστές προτάσεις σε αρκετά σημεία. Θεωρώ ότι οι άδειε απαιτούνται για αυτούς τους εργαζόμενους, τους χρειαζόμαστε επαναλαμβάνω και νομίζω ότι υποβάλλεται καλές σχετικά προτάσεις να δούμε και την κατοικία τους, το κατάλημά τους. Ε, θα χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες, ε, συμφωνώ με την κυρία Τούρουνεν, ε, πολλές φορές μένουν σε διαμερίσματα με τρομερά υψηλές τιμές που είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό της συνολικής αμοιβή του. Γι' αυτό λοιπόν πάνω στα σημεία αυτά συμφωνώ. Και Πιστεύω ότι το τρίτο μέρος θα πρέπει να διαγραφεί. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει ε, τα κοινωνικά επιδόματα, οτιδήποτε έχει με την κοινωνική ασφάλιση και για τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία χρειάζεται πραγματικά να ισχύσουν όσο γίνεται καλύτερα. Αλλά αυτό αποτελεί μια άλλη πρόταση διαφορετική από εκείνη με την οποία τώρα εμείς ασχολούμεθα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τις ε, συγκεκριμένες συνέπειες των όσων έχουν να κάνουν με εμάς, με τη δική μας την υπόθεση, το δικό μας το θέμα και σε ορισμένες ε, τρίτες χώρες ε, ε, ισχύουν πολλά και δύσκολα σε μερικούς τομείς και σίγουρα χρειάζεται ίση και δίκαιη αντιμετώπιση για αυτήν την εποχιακή εργασία να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η αυτό το διοικητικό βάρος και για τα εργατική ατυχήματα επίσης χρειάζεται να έχουν μια ασφάλεια. Τόμας και μετά Τόμας Μάν. Εδώ με τον κύριο Κοφεράτη σκοπεύουμε να συνεργαστούμε για να βρούμε λύσεις για τα πολύ ευάλωτα αυτά άτομα που πολύ συχνά είναι ε, αντικείμενο εκμετάλλευση. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή είναι σημαντική για να βελτιωθεί το κείμενο τη οδηγία. Υποβάλαμε τροπολογίες για το θέμα του ελέγχου. Είναι σημαντικό, εφόσον είδαμε να υπάρχουν ε, πολύ κακές κοινωνικές συνθήκες και αυτό από χρόνια, να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Η οδηγία αυτή αφορά την μετανάστευση μεν, αλλά πρέπει να σκεφτούμε το πεδίο αρμοδιοτήτων μας. Ε, η κυρία του των Πρασίνων το ανέφερε ήδη. Έχουμε εδώ κάποιες ε, συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά τις ε, γενικά ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει όσον αφορά τη, γενικά τη γενική εφαρμοσιμότητα των συλλογικών συμβάσεων ότι δεν είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τις διατάξεις των κρατών μελών αυτή η γενική, ο γενικά θεσμευτικός χαρακτήρας είναι κάτι που δεν τονίζεται εδώ επαρκώς και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες σχετικές προτάσεις και χαίρομαι που θα μπορέσουμε περαιτέρω να συζητήσουμε το θέμα με τους συζητητές. Μπορούμε νομίζω να βρούμε ένα πιο ακριβές σύστημα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τουρούνεν, ζητήσατε να παρέμβετε ξανά. Ναι, με συγχωρείτε. Θέλετε να αντιδράσετε σε όσα είπε η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Όχι, όχι, μια πολύ σύντομη διευκρίνηση την βρίσκω πολύ σημαντική. Έχουμε την τροπολογία 43, όπου λείπει ένας όρο και αλλάζει όλο το νόημα. Αυτό που θέλουμε να λέγεται ότι με την επιφύλαξη του γεγονότο ότι οι αρχέ αυτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να παρεκκλίνουμε από τι αρχέ για την ίση ε, πληρωμή, τι ίσε αποδοχέ και ε, τι ίσε συνθήκε εργασία. Ξεχάσαμε τέλο πάντων ε, μία λέξη και άλλαξε ολόκληρο το νόημα γιατί δεν αναφερόταν αυτό για παρέκκληση. προέδρο. μάλιστα. Θα γίνει διαφορετικό λοιπόν σημείωμα για τι τροπολογίε. Να προσταθεί αυτό που είπα. Το κύριος Μαν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι εδώ στην Επιτροπή μας για να πούμε όλοι μαζί ότι αυτό που θέλουμε είναι η ίση μεταχείριση. Δεν αφορά το θέμα μόνο τους υπηκός τρίτων χωρών, αλλά και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει η ίση μεταχείριση. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή αυτή θα βρούμε οπωσδήποτε με εκείνη θέση. Δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι πια στην παρανομία. Θα πρέπει να υπάρχουν οι διατάξεις που θα αναφέρουν αυτά που χρειάζονται, δηλαδή ασφάλεια, η δυνατότητα να, κάνουν αυτό που πρέπει στις εργασίες τους, να είναι σωστά, σωστή η όρη διαμονής τους. <clears throat> Γιατί συνήθως ε, μιλάμε για, την, ε, για τους όρους διαμονής μόνο όταν πάλι κάποια τηλεοπτικό σταθμό έχει ανακαλύψει αυτά που γίνονται και που είναι πραγματικά εξωφρενικά. Αλλά δεν θέλουμε να φτάνει εκεί. Θέλουμε ε, να είναι καλή όρη. Δηλαδή δεν αρκεί να του πούμε εντάξει σε λίγο χρονικό διάστημα θα κερδίσετε πάρα πολλά χρήματα, πολύ περισσότερο από το μπορούσατε να κερδίσετε στην ε, πατρίδα σα, αλλά με ποιου όρου. Γιατί υπάρχουν κάποιε οργανώσεις που του φέρνουν εδώ και ε, οι άνθρωποι είναι σαν, ε, σαν ε, φυλακισμένοι. Έχω έναν εδώ στην στους συνεργάτες μου αυτή τη στιγμή. Κάποιος που ήταν χωρίς ε, ε, υποκότα, εργάστηκε εδώ στο Βέλγο, στη συγκομιδή και στο τέλος δεν τον πληρώσαν καθόλου τίποτα, τίποτα, ούτε πεντάρα. Και του είπαν, πω, άμα δεν σ' αρέσει πήγαινε στο δικαστήριο να διαμαρτυρηθείς. Ο άνθρωπος δεν είχε κανένα δικαίωμα. Λοιπόν, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να βρούμε από κοινού μια σωστή προσέγγιση. Μου φαίνεται πάρα πολύ σωστό να πούμε θα πρέπει βέβαια να εμπλακούν και οι κοινωνικοί εταίροι. Θα πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να υπάρχει επιβολή κυρώσεων. Δεν μπορούμε να πούμε εντάξει δεν περάζει. Θα πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις που θα τηρούνται, που θα ελέγχονται και μόνο τότε έχουμε τη ε, δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους τρόπους αυτούς με αξιοπρέπεια. <coughs> Τέλος. Είχαμε για αρκετό καιρό την συζήτηση της διαφοροποίησης ανάμεσα στους εποχιακά εργαζόμενους και τους άλλους. Ε, υπάρχει στη Γεωργία όμως αυτό το θέμα των εποχιακά εργαζόμενων και άμα δούμε ε, ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε εντάξει, κερδίζουν κάποια χρήματα, μπορούν να διατηρήσουν στη ζωή στην ε, πατρίδα τους και γι' αυτό ξαναέρχονται και ξαναέρχονται χωρίς να διαμαρτυρηθούν, θα πρέπει να είμαστε εμείς κάποιος πιο λογικοί. Να ε, εμπλακούν και οι δύο πλευρές και τα δύο κράτη, και το, το κράτος προέλευσης και το κράτος υποδοχής. Σκιώδης ηγητής το είπε ξεκάθαρα ποια είναι η ευθύνη των κρατών μελών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κοινή πρωτοβουλία εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Κύριε Μπαλντασάρ, κάποιο άλλο συνάδελφος που θα επιθυμούσε να λάβει το λόγο. Όχι, ο κύριο Μπαλντασάρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή είναι η απαιτούμενη πρόταση. Έχουμε αυτή την πραγματικότητα της εποχιακής εργασίας επειδή δεν έχουμε τα κατάλληλα εργατικά χέρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί από αυτούς τους εποχιακούς εργαζόμενους ε, αντιμετωπίζουν ε, δυσμενείς συνθήκες, άσχημες συνθήκες, ε, τους εκμεταλλεύονται και πολλές φορές δεν σέβονται οι εργοδότες και τον νόμο. Γι' αυτό θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια κατάλληλη ρύθμιση στη γεωργία, στα αποκρεπευτικά, στον τουρισμό. Εκεί κυρίως εργάζονται τα άτομα αυτά και εκεί προσλαμβάνουν ακριβώς ε, εργατικά χέρια από τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι ο Σέρτζιο θα επιτελέσει άριστο έργο γιατί τα σημαντικά, τα κύρια θέματα έτσι κι αλλιώς ε, τα βλέπουμε όλοι με τον ίδιο περίπου τρόπο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορούν να εφαρμόσουν ένα κριτήριο που να εφαρμόσει ότι η κενή αυτή θέση δεν μπορεί να πληρωθεί από ντόπια εργατικά χέρια σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να προστατευθούν όπως πρέπει τα δικαιώματα αυτών των εποχιακά εργαζομένων ή σε αντιμετώπιση με τους ε, πολίτες ε, των ε, κρατών μελών. Βέβαια, σε αυτή την εποχή πρέπει να περισσουμε το κόστος. Αλλά τι γίνεται, θα πρέπει να δούμε βέβαια και την παγκοσμιοποίηση, αλλά όχι όμως με ε, κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επίσης, οι συλλογικέ συμβάσει θα πρέπει να σεβαστές από παντού στην χώρα αυτή παντού και σε βιομηχανικό επίπεδο κλπ. Και θα πρέπει να συμφωνούν με την εθνική πρακτική και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίζει τη φύση και τη διάρκεια αυτής της εποχιακής εργασίας ανάλογα με τις απαιτήσει της και τα χαρακτηριστικά της και κάτι ακόμα θα πρέπει να εγγυηθούμε σε αυτούς τους εποχιακά εργαζόμενους ένα κατάλημα κατάλληλο ε, που να μην είναι πολύ πιο ακριβό από το κανονικό, ε, να μην αποτελεί μεγάλο μέρος του μισθού τους, της αμοιβή τους. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε μια πολύ σωστή δουλειά για μια έκθεση που ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των εργαζομένων αυτών, αλλά και των, των χωρών μας. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Τώρα κάποιος άλλος συνάδελφος θα επιθυμούσε το λόγο. Όχι. Η Επιτροπή, κυρία Σμιτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ζητήσω συγγνώμη Βρισκόμουν σε άλλη συνάντηση, γι' αυτό καθυστέρησα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μερικές παρατηρήσεις μετά τη συζήτηση που έγινε και για τις τροπολογίες που αποβλήθηκαν. Να πω ότι έγινε σαφές από τη συζήτηση ότι στόχος της, προστασί... της πρότασής μας είναι να έχουμε ευέλικτο σύστημα υποδοχής ώστε να μπορέσουν οι επίκοτροι των χωρών που εργάζονται σε εποχικοί εργαζόμενοι να φτάνουν και να είναι διαθέσιμοι γρήγορα όταν χρειάζονται. Αυτό βέβαια όχι εις βάρος των Ευρωπαίων Επικών. Γι' αυτό η πρότασή μας προβλέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν τα δικά τους τεστ για τις αγορές εργασίας τους και να φροντίζουν και οι δικοί του υπήκοοι να γίνονται αποδεκτοί ω εποχικοί εργαζόμενοι. Κάτι σημαντικό που αναφέρθηκε στην εδώ συζήτηση είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τι καταχρήσει του συστήματο. Δηλαδή, σημαντικό θα είναι να προβλεφθούν και κυρώσει και τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν τι απαραίτητε επιθεωρήσει και ελέγχου. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε βέβαια και περιττή γραφειοκρατία εδώ. Κατά τα άλλα πρόταση αυτή θέλει να καλύψει και τους εργαζομένους με χαμηλές δεξιότητες ε, και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια ευάλωτη ομάδα εργαζομένων και πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες ακριβώς που έχουν υποβληθεί μπορούν να ενισχύσουν το στοιχείο της προστασίας και της δικής μας πρότασης. Θα έχουμε νομίζω λοιπόν την ευκαιρία να επανέλθουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξυπηρετήσει για να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση και να προστατεύεται και αυτή η κατηγορία εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα που προβλέπονται, όταν σχεδιάσαμε την πρότασή μας, θέλαμε να διασφαλίσουμε ίση μεταχείριση. Οι εργοδότες που απασχολούν υπηκόστοι των χωρών να διατηρούν το ανταγωνιστικό του δικαίωμα, αλλά να υπάρχει και συνέπεια μεταξύ του κεκτημένου μα στον τομέα τη νόμιμη μετανάστευση. Ε, ήμουν στην Επιτροπή Λίμπε συγκεκριμένα προηγουμένω, γι' αυτό και καθυστέρησα και ακριβώ κάποια στοιχεία του κειμένου αυτού συζητήθηκαν. Ε, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Βεβαίω η κατάσταση δεν είναι ακριβώς η ίδια σε σχέση με, με το μεταναστευτικό πακέτο γενικότερα, γιατί εδώ μιλάμε για εποχικού εργαζομένου, που έρχονται προσωρινά, για μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ακριβώς υποβάλαμε και την πρότασή μα. για να λάβουμε υπόψη τον προσωρινό χαρακτήρα τη παραμονή. Σε ό,τι αφορά την ίση λοιπόν μεταχείριση, Τη συνδέσαμε με μια σειρά από δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, της ε, συμμετοχής σε συντεξιωτικό ταμείο. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρει κάτι και ο συνάδελφος. Εδώ την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δεν προβλέψαμε κάτι ιδιαίτερο για την εκπαίδευση βέβαια. Λόγω ακριβώς της προσωρινής παραμονής των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας, πράγματι προτείναμε ίσο επίπεδο δικαιωμάτων όπως με τους ε, ε, σε μετάθεση εργαζομένων τη ίδια ε, τη Ευρωπαϊκή Ακόμα και αν η κατάσταση των αποσπασμένων εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάτω μέλος σε κάτω μέλος είναι διαφορετική γιατί εκεί υπάρχει σύμβαση που διέπει την απασχόλησή τους, θέλαμε να μην δημιουργηθεί μια ξεχωριστή τελείως κατηγορία. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως η νομική προστασία των εργαζομένων στο κείμενο. Επίσης προβλέψαμε ένα ισότιμο επίπεδο διαβίωση χωρί να προκαθορίζουμε όμω τι ακριβώ θα πει αυτό. Δεν υπάρχει σχετικό ορισμό. Τα κάθε μέρη λοιπόν θα πρέπει να προβλέψουν κάποια πρότυπα σε ό,τι αφορά την υγιεινή του περιβάλλοντο τι ελάχιστε συνθήκε καλή διαβίωση και βεβαίω κάποια κατευθυντήρια κάποια κατεύθυνση την έχουμε από το κεκτημένο μας με τις μακράς διάρκειας παραμονές και την οικογενειακή πανένωση. Οι καλέ συνθήκε λοιπόν διαβίωση από εκείνα τα κείμενα μπορούν να μα εμπνεύσουν για να πετύχουμε περισσότερη σαφήνεια στο τι εννοούμε εδώ. Οι κυρώσει επίση είναι σημαντικέ. Θα το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Έχουμε οδηγία για τι κυρώσει κατά των εργοδοτών που παρανόμως απασχολούν επικόστρια των χωρών. Η οδηγία αυτή θα τεθεί σε ισχύ στις 20 του Ιούλη, συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώ η κατάσταση τη μεταφορά βέβαια τη οδηγία αυτή δεν είναι ιδανική προ στιγμήν. Οπότε βάσει τη συνθήκη η Επιτροπή θα κινήσει τι απαραίτητε διαδικασίε κατά των κατομελών που δεν έχουν υλοποιήσει την οδηγία. Δεν την έχουν μάλλον μεταφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη διασύνδεση τη εν λόγω πρόταση με την ε, οδηγία για τι κυρώσει. Διότι είναι πολλοί οι παρανόμω διαμένοντε που εργάζονται σε πολλού τομεί. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ. Και αν κανείς άλλος δεν επιθυμεί το λόγο, τότε ο εισηγητής μας. Και πάλι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, όλους για τις παρατηρήσεις τους που θα μας βοηθήσει στην εργασία μας. Να καθησυχάσω την συνάδελφο του Ρούνεν ε, Πολύ καλά κατάλαβα ότι στην 53 τροπολογία υπήρχε ένα λάθος γιατί θα μας εξέπλησε διαφορετικά μια αλλαγή στάσης από πλευρά των πρασίνων. Εντάξει, άρα λοιπόν το έχουμε κατανοήσει. Δύο παρατηρήσεις γρήγορα γρήγορα μετά από όσα άκουσα. Αυτός ο στόχος που όλοι συμμερίζονται κατά την απόψή μου έχει να κάνει με ένα μέτρο που να είναι αποτελεσματικό σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς στις όλες δραστηριότητες στην εργασία. Και ιστορικά στον τομέα αυτό εκεί διαπράττονται οι χειρότερες αδικίες και άνδρες γυναίκες όσοι εργάζονται εκεί αντιμετωπίζουν συνθήκες εργασίες που μερικές φορές είναι και απάνθρωπες. Ας πούμε το τι συνέβη στη χώρα μου, την Ιταλία, με το Ρεζάρνο, με εδώ και το κοινοβούλιο μας ασχολήθηκε επί μακρόν. Ρύθμιση λοιπόν με το κριτήριο της ίσης αντιμετώπισης των ίσων δικαιωμάτων, κάτι τέτοιο είναι σημαντικό και αυτό για μια κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά επίσης και για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις γιατί αποκλεί οποιαδήποτε δυνατότητα dumping και έτσι έχουμε ακριβώ τις ίδιες δυνατότητες σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον, ε, κάτι το γενικό, η οδηγία τους πιο εκτεθειμένους, τους ασθενέστερους βοηθάει, αλλά ταυτόχρονα ρυθμίζει την αγορά τα πράγματα για τις επιχειρήσεις, γιατί μειώνει τις δυνατότητες dumping. Και ακόμα βέβαια η ευλογιστία και η ευκαμψία θα πρέπει να ισχύουν. Εδώ μιλάμε για συνθήκες που έχουν να κάνουν ας πούμε όπως την συλλογική σύμβαση, την κοινωνική προστασία που διαφέρουν από τη μία χώρα κάπως ε, στην άλλη αλλά χρειάζεται ένας ενιαίος χαρακτήρας αντιμετώπισης και επακριβώς να διευκρινίσουμε τι ακριβώς ε, πρέπει μπορούν να κάνουν τα άτομα αυτά και για να διευκρινίσω καλύτερα και την απόψή μου. Όταν λέμε ότι οι εξαιρεσει θα πρέπει να προβλέπονται από τα κράτη-μέλη στη συνοήση με τους κοινωνικούς εταίρους δεν ξεχνάω ότι ο νόμος θα είναι η τεχνική λύση και τα κοινοβούλια θεσπίζουν τους νόμους, αλλά μπορούν καμιά φορά να το κάνουν αγνώντας τους κοινωνικούς εταίρους, είτε θεσπίζουν νόμους βάσει μιας στενής σχέσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό το τελευταίο είναι και ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Κάτι ακόμα για το κατάλημα. Μιλάμε για κόσμο που έρχεται από μακριά και δεν έχουν την ίδια δίκαιη σχέση με τον κόσμο γύρω τους. Από τη στιγμή που ψάχνουν για ένα κατάλημα ε, δεν έχουν ε, τους κατάλληλους τρόπους, τα κατάλληλα μέσα για να επιλέξουν την καλύτερη λύση όπως θα μπορούσε να το κάνει κάποιος πολίτης που εκεί είναι, εκεί ζει εδώ και αρκετά χρόνια. Σε αυτό, θα πρέπει να προσέξουμε και να βρούμε και λύσεις που θα τους βοηθήσουν για να μην επιβαρύνονται. Και η τάση είναι να ζουν μαζί και οι εταιρείε αρκετές φορές ε, ευνοήθηκαν από αυτό, εποφελήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα συγκεκριμένοι στον ορισμό τι σημαίνει αξιοπρεπές κατάλημα, ώστε να τους εξασφαλίσουμε εκείνο το χρονικό διάστημα που μένουν μαζί μας να κατοικούν όπως πρέπει. Και κοινωνική δικαιοσύνη λοιπόν. Αυτά θα τα δούμε και τις λεπτομέρειε τις μέρες που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λέει πρόεδρος ε, να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι ε, αρκετές ε, τροπολογίες κρίθηκαν ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν εδώ γιατί δεν είναι αρμόδια αρμοδιότητες δικές μας και θα σας ανακοινώσουμε το σχετικό κατάλογο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τώρα, μετά από την συζήτηση αυτή, θα προτείνει συμβαστικές τροπολογίες ο εισηγητής και εμείς θα τις συζητήσουμε τις 19 Σεπτεμβρίου και βέβαια θα ψηφίσουμε τις 6 Οκτωβρίου και η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών το Νοέμβριο θα αποφανθεί τελικά. Ε, είμαστε στο σημείο 16 τώρα της ημερησίας διάταξης. Δεν έχει μάλλον έχει αρκετή σχέση με το σημείο που μόλις συζητήσαμε, δηλαδή έκθεση της κυρίας Γιακονσάρη για προποθέσεις εισόδου και διαμονής επικών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης. Ο κύριος Σέρκας θα την αντικαταστήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγγήτριά μας δυστυχώς Ακριβώς ε, δεν μπορεί να είναι μαζί μας ε, κυρία Μαλγκοζάτα Χάντζικ ε, και με ενημέρωσε σχετικά με την έκθεση αυτή και ελπίζω να σας πω ακριβώς πως έχει κατάσταση. Ήδη γνωρίζετε το προσχέδιο και τις τροπολογίες και έχουμε 167 τροπολογίες εκτός από τις δικές της. Τα πρώτα για τα οποία με ενημέρωσε είναι ότι ουσιαστικά αυτά τα σημεία, τα κύρια συζήτησης ε, έχουν καθοριστεί επακριβώς και ανάμεσά μας ε, υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη σύνταξη μιας έκθεσης όπου τα κύρια σημεία μπορούν να μας δουν αρκετά σύμφωνος. Βέβαια όλοι μας ξεκινάμε από μια πραγματικότητα ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική οδηγία τώρα που βλέπουμε τον παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τις πολυεθνικές κλπ. και χρειάζονται ρυθμίσεις όλα αυτά για να είναι περισσότερο ευλίγιστα και εύκαμπτα για την εργασία, ή για την απασχόληση του προσωπικού αλλά αυτή τη στιγμή που έχουμε περισσότερη κινητικότητα και θα έλθουν ακόμα περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστούν, θα πρέπει ιδιαίτερα με ακρίβεια να δούμε μερικά θέματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων που είναι ήδη εδώ και που εκείνων που έρχονται, που δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι μεν ή οι δε περισσότερο από τους άλλους. Και επίσης επειδή Έχω, δεν έχουμε σύνορα στην εσωτερική αγορά, βλέπουμε ακριβώ πώ έχει κατάσταση, θα πρέπει να υπάρχουν τα ελάχιστα απαραίτητα που θα βοηθήσουμε την ε, ανταγωνισμό ανάμεσα σε εταιρείε, όχι ανάμεσα στα κράτη. Να αποφύγουμε το dumping το κοινωνικό του ενός κράτους απέναντι στο άλλο και να υπάρχουν οι ελάχιστε κοινωνικέ ρυθμίσει που να καλύπτονται από την οδηγία. Βλέπουμε πως πρέπει να έχει αυτή η οδηγία και μπορούμε τώρα που λέμε καλύτερη ρύθμιση και νομοθεσία να έχουμε ακριβώ μια σαφή, συγκεκριμένη, διάφανη νομοθεσία και να μην υπάρχουν ασάφειες. Αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα δεινά προβλήματα που έχουν να κάνουν με κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνδικάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αντιμετωπίζουν διαφορετική οδηγία που στο κοινωτικό επίπεδο ρύθμιζε τα πράγματα σχετικά με τους μετακινούμενους εργαζόμενους. Βλέπουμε ανεπάρκειες, ότι, δεν υπάρχουν, ότι υπάρχουν ασάφειες, υπάρχει μια σύγχυση μεθοδολογική, αντιφατική νομοθεσία και εδώ. Μας οδήγησαν όλα αυτά σε ένα χάος, σε αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Θα πρέπει η οδηγία αυτή, η οποία και θα ρυθμίσει την κινητικότητα των εργαζομένων εκτός κοινότητας, να μην έχει να κάνει μόνο με τη φιλοσοφία και τις παραμέτρους της σημερινής οδηγίας, γιατί τότε θα πολλαπλασιαστούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Και υπάρχουν Τρία δισεκατομμύρια εργαζομένων παντού γύρω και που θα πρέπει να δούμε την πρώτη προσέγγιση και να ακούσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που είναι εδώ μαζί μας πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτής της καταστάσεως και να μην είμαστε πολύ συντηρητικοί θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με αυτήν την οδηγία, την οδηγία μετακίνησης. Η Επιτροπή λέει ότι χρειάζεται μια τρομερή προσπάθεια για την εναρμόνιση και το συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρυθμιστικά την απόψή μας θα πρέπει να δούμε και την τοποθέτηση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να βελτίωθει η οδηγία για την ε, μετακίνηση των εργαζομένων ε, μέσω ρυθμίσεων που να συμφωνήσουν 27 κρατη να δούμε τις μεταφράσεις εγγράφων, όλα αυτά και υπάρχουν ε, τρομερά πράγματα που πρέπει να γίνουν, πολλή δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ίδια θα συμβαίνουν και σε πολλές χώρες και ότι θα μπερδέψουμε και άλλους αν έχουμε ασάφειες. Θα πρέπει κανονικά να λύσουμε προβλήματα που δεν έχουν λύσει οι νομοθέτες. Ε, καλύπτει όλους αυτή η ιδέα ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στη σημερινή πραγματικότητα, όπως επίσης και σαν και όχι έτσι να ενεργούμε από κεκτημένη ταχύτητα με τις ίδιες ανυπάρκειες, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινοτικοί εργαζόμενοι. Αυτό. Να δούμε και για την Λίζα Λιακονσάρη τι αναφέρει σαν τρία κύρια σημεία και να σας πω ότι προετοιμάζεται για να πετύχει συμβαστικές λύσεις, να υπάρχει μια ικανοποιητική βάση για όλα αυτά. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε αρκετά σημεία όπως το σημείο εφαρμογής της οδηγίας. Μετά από την ανάγνωση αυτών των 170 περίπου τροπολιών θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε μια ευρεία πλειοψηφία για να δούμε πέρα από την εποχιακά εργαζόμενος και να μην μπερδέψουμε τη μία οδηγία με την άλλη, να είναι μια έργας, μια οδηγία για εκείνους που έχουν έδρα σε άλλες χώρες, αλλά μην τον μπερδέψουμε με την εποχιακή εργασία. Παραλαμβάνω υπάρχει μια πλατιά βάση για να συμφωνήσουμε και να αποκλείσουμε τον κατασκευαστικό τομέα και αρκετές τροπολογίες μας επιτρέπουν τα κράτη-μέλη με τους κοινωνικούς εταίρους να μπορέσουν να δουν ποιος, ποιο είναι το σημείο το πεδίο εφαρμογής περισσότερο περιοριστικό και από τη στιγμή που θα υπάρξει μια συμφωνία. Άλλο πρόβλημα, οι ορισμοί. Γιατί εδώ σε μια οδηγία που θα πρέπει να ανοίξει του δρόμου για άτομα με δεξιότητες στις πολυεθνικές εταιρείες και είναι ένας, ε, τι είναι ένας μάνατζερ, τι είναι ένας ειδικός, θα πρέπει να το πούμε επακριβώς και τι είναι κάποιος που ασκείται, κάνει την πρακτική του υπό τις συνθήκες αυτές και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες, σε αυτές τις επιχειρήσεις και αρκετές τροπολογίες αρκετά ενδεικτικές από διάφορες ομάδες που ζητείται ένας κατάλληλος ορισμός. Να λέει ότι κάποιος που μετακινείται ε, Βέβαια υπάρχει μια αρχαιότητα αλλά να μην καταστατηγείται το πνεύμα της οδηγίας και να έχουμε από την άλλη μεριά ε, εργαζόμενους που να προσλαμβάνονται μόνο και μόνο για να αποσταλούν στην Ευρώπη, αλλά να υπάρχει μια κάποια αρχαιότητα που να αναγνωρίζεται σε αυτούς και θα πρέπει ας πούμε να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όπως έξι μήνες που να έχουν προσδειχθεί πριν και άλλοι που λένε περισσότερο. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ οι τροπολογίες αυτές ε, σαν Χέντελ, διάφοροι ορισμοί με το 96 τροπολογία Χέντελ, 90 επίσης, 89 Χίρς, 82 επίσης ε, που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ολοκληρώνω εδώ. Τη στιγμή που πρόκειται για μια οδηγία στην οποία μιλάμε για εργαζόμενους με δεξιότητες ε, και έχουμε μια κάποια έννοια με ισχυρή βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ισχύουμε ακόμα περισσότερο. Μια σωστή αναφορά θα ήταν η οδηγία που, ναι, που έχει προετοιμαστεί από άτομα με προσόντα, με δεξιότητες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις συμβαστικές λύσεις για να προσεγγίσουμε τους ορισμούς που ισχύουν ήδη στο Μπλούκα στην οδηγία αυτή. για την, ε, για την μπλε κάρτα λοιπόν. Αυτά. υποστηρίζουμε την εισηγήτρια. Έχουμε 172-173 Ρενσούλη Μπαλτασάρ και άλλων Χέντελ, α πούμε, Λάμπερτ, 169-173 Σρέντερ, ε, σοσιαλιστέ, διάφορε τροπολογίε και νομίζουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πλειοψηφία γύρω από όλα αυτά και που αναφέραμε όπω και για του εποχιακά εργαζόμενου. Αυτό έχει τρομερή σημασία να δούμε ακριβώ αυτό το κριτήριο ε, ότι όποιο έρχεται στην Ευρώπη πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με του Ευρωπαίου εργαζόμενους. Όχι να αντιμετωπίζεται χειρότερα, δυσμενέστερα από αυτού, Λοιπόν, ε, ισότητα δικαιωμάτων ε, και για τη εργασία, για την κοινωνική προστασία. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε έτσι την ε, δομέα της εργασίας και να αντιμετωπίζονται χειρότερα από τους Ευρωπαίους εργαζόμενους οι υπόλοιποι γιατί δεν στέκει με τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χάρτα θεμελιών δικαιωμάτων και με τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να υπάρξει μια ηθική που να ισχύει σεβόμαστε όλους χωρίς διακρίσεις δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις η ε, βάρος αυτών και θα ήταν τρομερά λάθο να έρχεται εδώ κόσμο στην Ευρώπη κατά από δυσμενέστερες συνθήκε, γιατί έτσι καταστρέφεται ο κοινωνικός ιστός, η εμπιστοσύνη των εργαζομένων, η αλληλεγγύη μεταξύ τους και δημιουργείται και η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Δεν μπορούν να έρχονται εδώ στην Ευρώπη με λιγότερα δικαιώματα πως εδώ εργάζονται. Με τη διαλογική οι Ευρωπαίοι ακριβώς εργαζόμενοι καταλαβαίνουμε γιατί διαμαρτύρονται γι' αυτό και δεν δέχονται αυτή την άδικη κατάσταση χωρίς καμία, καμία λογική. Και τώρα που το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο συζητάμε για το τι ακριβώς κάνουμε και λέμε ότι είμαστε στην πρωτοπορία κατά οποιασδήποτε διάκριση Σίγουρα οποιαδήποτε μορφή διάκριση σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί και να μην ισχύσει. Αγαπητοί, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική οδηγία, τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας, οι εταιρείες μας. Δεν θα πρέπει να κάνουμε λάθος στην αντιμετώπιση αυτών των εργαζομένων. Έτσι, γιατί εάν ε, παρεκκλίνουμε, όπως είπε ο Νάλφος, θα μπούμε σε ένα δρόμο γεμάτο ε, προβλήματα θα παρεκκλίνουμε από την ιδέα της Ευρώπης κατά των όσων ισχύουν που είναι τα σωστά για εκατομμύρια εργαζόμενους εδώ τη στιγμή που θα πρέπει να έχουμε μια εσωτερική αγορά με αρχές, με αξίες, μια εσωτερική αγορά όπου ε, διαφορετικά θα έχουμε τη διαφθορά, τα προβλήματα, τα σταλίες, όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με τους κοινωνικούς εταίρους και να καταλάβουμε ότι όποιος έρθει θα πρέπει να σωματώνεται στο πρότυπα και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όχι απλά και μόνο να δημιουργήσουμε ένα κενό στην όλη μας ρύθμιση. Είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν άλλωστε στα κράτη μας μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Διεξοδικότατη ήταν. Αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία και αυτή η συζήτηση, κυρία Εσάγια και μετά η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη και για αυτή την οδηγία, όπως και για την προηγούμενη. Να θυμίσω όμως ότι το πεδίο της οδηγίας αυτής είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Στον τομέα ICT έχουν υψηλά προσόντα, δεξιότητες υψηλού επίπεδου, οπότε δεν έχουμε τα φαινόμενα εκμετάλλευσης ίσως και καταχρήσεων που αναφέραμε προηγουμένως σε σχέση με την με τους εποχικούς εργαζομένους. Πραγματικά όμως, πάλι και εδώ οφείλουμε να είμαστε σαφέστατοι στου ορισμούς, όπως είπε και ο κύριος Σέρκας. Ένα από τα παραπλανητικά ζητήματα εδώ είναι να βρούμε τον τρόπο που θα διασυνδέσουμε αυτή την οδηγία με την οδηγία για την μετάθεση των εργαζομένων. Το στοιχείο αυτό το έθιξε και ο κύριος Σέρκας. Εάν εξαλείψουμε όλες τις αναφορές στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, τη μετάθεση μάλλον των εργαζομένων, όπως έκανε η κυρία Γιάκοντσαρη, δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ο καλύτερος τρόπος και θα διευκολύνουμε τα πράγματα. Πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τι λύση θα προκρίνουμε. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι και αυτοί οι εργαζόμενοι εξορισμού είναι μετατιθέμενοι. Έχουν εργασιακή σύμβαση στις τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται. Οπότε πραγματικά είναι αποσπασμένοι, δηλαδή μετατεθειμένοι από τις χώρες αυτές. Πάντως, εάν το συζητήσουμε και με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, φαντάζομαι ότι τον σωστό συσχετισμό θα τον βρούμε θα τον αναφέρουμε ή θα τον εξαλείψουμε, πάντως μια σωστή διατύπωση θα τη βρούμε. Για τους ορισμούς τώρα, στο άρθρο 3, θα πρέπει να συναδούν με τις ε, διατάξεις της Συμφωνίας ΓΚΑΤ και θα πρέπει να αποσαφινιστούν επαρκώς ώστε να υπάρχει καλύτερος εντοπισμός των κατηγοριών που καλύπτονται από τις μεταθέσεις. Να αποσαφηνίσω και μια της δικές μου τροπολογίες, την 113, διότι ζητώ διαγραφή, πλήρη διαγραφή του κειμένου της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ορίσει συλλογικός μάλλον ε, ε, οικομενικώς εννοούμενες, ε, συλλογικές συμφωνίες στο κείμενο της Επιτροπής όμως ο ορισμός δίνεται έτσι που αντιφάσκει με την εθνική νομοθεσία τις εθνικές πρακτικές που έχουν επικρατήσει. Λόγου χάρη στις σκανδιναβικές χώρες οι ορισμοί, οι συμφωνίες μάλλον αυτές, οι συλλογικές συμφωνίες γίνονται από τους ε, εργαζομένους που εκπροσωπούνται από τις ε, συνδικαλιστικές τους οργανώσεις του κοινωνικού δηλαδή εταίρου, σε συνεργασία με του εργοδότε, τι ενώσει εργοδοτών. Εάν τώρα θέλουμε να επηρεάσουμε αυτού του ορισμού, θα είναι πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσουμε σε εθνικό επίπεδο. Σε χώρε όπου ήδη προβλέπονται σχετικοί κανόνε. Υπάρχουν δηλαδή συλλογικέ συμφωνίε. Ο ορισμό που τώρα προτείνεται διαφέρει από τα όσα ισχύουν σε εμά. Επίση, το θέμα της κοινωνικής ε, ασφάλισης. Αυτό που και ο κύριος Έρκας έφυξε. Εδώ έχουμε παρόμοιες ανησυχίες με αυτές που είχαμε όταν εξετάζαμε την οδηγία για την ενιαία άδεια. Η ίση μεταχείριση στο άρθρο 14 που να ορίζεται έτσι, ώστε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που βασίζονται στον, ε, στη χώρα εγκατάστασης να μπορούν να ακολουθούν τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας των ε, συστημάτων. Και αυτό γιατί στην κοινωνική ασφάλιση δεν έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις οδηγίες αυτές βλέπουν μια σειρά προβληματισμών σε σχέση με την κοινωνική ασφάλεια και την νομοθεσία της. Ανοίγονται θέματα που φύγουν τα κράτη-μέλη κατά τρόπο άστοχο. Ελπίζω λοιπόν να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα που τα αντιμετωπίσαμε και να την οδηγεί για την ενιαία άδεια. Επίση, θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσει όπου ένα εργαζόμενο καλύπτεται από δύο νομικά συστήματα ταυτόχρονα και πληρώνει φορέ και στα δύο. Και το κράτο μέλο δηλαδή, όπου βρίσκεται, και την τρίτη χώρα από που προέρχεται. Αυτέ μάλλον είναι οι βασικέ μα ε, ανησυχίε. Αυτά που τουλάχιστον ήθελα τώρα να θίξω υπολογίζω στην καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής και με τον εισηγητή και με τους άλλους σκεώδεις και στην καλή συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Πιστεύω ότι το κείμενο θα γίνει σαφέστερο και περισσότερο κατανοητό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χίρς και κυρία Σρέτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξ ονόματο των φιλελευθερών έχω να πω ότι και η οδηγία αυτή και οι τροπολογίες γενικά κινούνται προ σωστή κατεύθυνση. Αυτό που αναφέρθηκε συγκεκριμένα είναι ότι θα πρέπει να εξε... ότι εξαιρούνται εκείνοι που εργάζονται στι οικοδομές. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Αυτό που είναι μια αδυναμία και έχουμε υποβάλει σχετικές τροπολογίες είναι ο τομέας των ορισμών για να είμαστε αφενός σαφέστεροι και αφετέρου να μπορέσουμε να διασπάσουμε τους πολύ στενούς ορισμούς ούτως ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα ελιγμού εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή δεν πρέπει να αναφερόμαστε για αποφύρους πανεπιστημίων ή, ή ιδιαίτερα ε, άτομα με ιδιαίτερα προσόντα. Αλλά θα πρέπει να αφήσουμε ένα πολύ πιο γενικό ορισμό, ειδικευμένοι εργαζόμενοι κατά κάποιον τρόπο. Και κάτι άλλο. Τι είναι ένας όμιλος, τι είναι... Πώς υπάρχει δηλαδή ο συσχετισμός ανάμεσα στα διάφορα τμήματα μιας εταιρείας μιας μεγάλης εταιρείας. Και αυτό θα πρέπει να το ορίσουμε. Και έχουμε υποβάλει και κάποια άλλη τροπολογία όσον αφορά την ε, διάρκεια του χρόνου κατά το οποίο κάποιος ε, μπορεί να είναι μέλος αυτής της επιχείρησης. 12 μήνες λέγεται τώρα αυτό τώρα δεν είναι πια σύμφωνο με την πραγματικότητα του επιχειρησιακού κόσμου, ότι κάποιος θα πρέπει δηλαδή να είναι 12 χρόνια μόνιμο σε μια επιχείρηση για να μπορεί να αποσταλεί κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να μειώσουμε στους 6 μήνες είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Και ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό και για την γραφειοκρατική πτυχή θα πρέπει να είναι δυνατότητα για τα άτομα αυτά να μπορούν να εργαστούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Γιατί πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν, ας πούμε, ε, μία θεατρική στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην ε, Αγγλία και θα πρέπει παντού να μπορούν να εργαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να, πρέπει, να μην πρέπει να έχουν ειδική άδεια κάθε φορά. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το προβλέψουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Πάντως ε, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή λύση και θα ε, έχουμε τελικά ένα κείμενο που να αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σφέτερ και η μετά η κυρία Ισλόβισκια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκείνοι που ασχολήθηκαν εις βάθος με την οδηγία καταλαβαίνουν πόσες αντιφάσεις υπάρχουν μεταξύ εκείνων που πήραν το λόγο. Εμείς οι πράσινοι ασχοληθήκαμε εις βάθος με την πρόταση και υποβάλαμε τροπολογίες για σημαντικά θέματα σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν ιδίω ε, όσον αφορά τη νομική βάση. Δεν συμφωνούμε όμως με την εισηγήτρια που λέει ότι θα πρέπει η νομική βάση να είναι σύμφωνη με το εργασιακό δίκαιο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μετανάστευση και εκεί θα πρέπει να παραμείνει. Από την άλλη μεριά όμως αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για αποστολή. Γιατί αποστολή σύμφωνα με τη συνθήκη είναι μέσα στο τομέα της ελεύθερης προσφοράς υπηρεσιών. Εμείς ε, θέλουμε να είμαστε στην ελευθερική κίνηση των ατόμων και να παραμείνουμε στην δέσμη μετανάστευσης. Και αυτό έχει νόημα, γιατί αν κοιτάξει κανένας την οδηγία για τους ε, απεσταλμένους ή αποσπασθέντες, βλέπουμε ότι αυτή η οδηγία καλύπτει τα άτομα αυτά από τρίτες χώρες. Δεν χρειαζόμαστε νέους κανόνες. Εάν πρόκειται για απόσπαση από τρίτη χώρα, ισχύει αμέσως η σχετική οδηγία. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Και γι' αυτό η Κομισιόν προσπάθησε σε αυτό το φάκελο να κάνει μια διάκριση, αλλά δεν το έκανα με αρκετή σαφήνεια. Και αυτό, από όσο κατάλαβα εγώ, οφείλεται στο γεγονός ότι το ε, Συμβούλιο θεωρεί ότι πρόκειται για απόσπαση και όχι για μετακίνηση ατόμων, γιατί υπάρχει συνθήκη. Και η μετανάστευση βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη μετακίνηση ατόμων και όχι στην προσφορά υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα πρέπει να κινηθούμε στο πυλώνα που αφορά την κίνηση των ατόμων και όχι στον πυλώνα που αφορά τις υπηρεσίες. Αυτό που πετυχαίνουμε εμείς δηλαδή με τις στροπολογία μας είναι πιο αυστηρή διάκριση μεταξύ εκείνων που είναι σαφή ούτως ή άλλως, δηλαδή αν κάποιοι έρχονται εδώ μέσα στα πλαίσια μας απόσπασης, καλύπτονται από την οδηγία της υπηρεσία, το έχουμε πει αυτό, ή είχε διακανονιστεί. Αν όμως έχουμε αυτά τα άτομα εδώ, έρχονται σαν εργαζόμενοι. Και μάνατζερ να είναι πάλι είναι στο κάτω-κάτω. Έρχονται δηλαδή σαν μεμονωμένα άτομα τα οποία κινούνται μέσα στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης από τη μία θηγατρική στην άλλη της ίδιας επιχείρησης. Και αυτό έχει δίκιο το Συμβούλιο ότι αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα της Στοκόλμης. Παραμένει μέσα στην ελεύθερη διακίνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι κάποιος δεν πρέπει να ζητάει κάθε φορά ειδική άδεια. Αυτά είναι σαφή. Αυτό που ήθελε η Κομισιόν ήταν ότι κάποιος που μέσα στα πλαίσια μας επιχείρηση πάει από τη μία χώρα στην άλλη δεν πρέπει να αρχίζει πάντα από το μηδέν, σαν μόνος έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι σαφές γιατί αυτό πρέπει να καταλογιστεί μέσα στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Και δυστυχώς οι μεγαλύτερες αντιδράσεις θα είναι στο Συμβούλιο που θα πούνε ακόμα και αν υπάρχει μία σύμβαση εργασία σε τρίτη χώρα, έχουμε εδώ την ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτή είναι η βάση και για τις επιχειρήσεις. Να μπορούν να μεταφέρουν, να μετατοπίσουν, να αποσπάσουν τους εργαζόμενους τους από τη μία τη στην άλλη. Το πρόβλημα που δεν λύνεται από την Κομισιόν είναι εκείνα τα άτομα που έχουν μια συμβασία εργασίας και που υπόκεινται στην, ε, στις διατάξεις της ελεύθερης κυκλοφορίας. Και γι' αυτό δεν συμφωνούμε με τους σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι είναι θέμα εργασιακού δικαίου, αλλά είναι θέμα μετανάστευσης κατά τη γνώμη μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξεκάθαρο διαχωρισμό από την οδηγία απόσπασης. Γι' αυτό το αντιστρέψουμε. Είναι πιο απλό και για τις ε, επιχειρήσεις ότι αν πρόκειται για απόσπαση δεν υπάγεται σε αυτή την οδηγία. Απ' την άλλη μεριά χρειαζόμαστε ειδικέ εξαιρήσεις για τον τομέα των οικοδομών. Γιατί εκεί έχουμε πάντα μια προσφορά υπηρεσίας. Και έχουμε τη στήριξη της και δεν συζητιέται καν ότι είναι θέμα προσφοράς υπηρεσίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ορισμό για τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγίας και θα πρέπει να πούμε ότι είναι άτομα με υψηλά επαγγελματικά προσόντα. Πρέπει να το πούμε σε κάθαρα γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια ανάμειξη και είμαστε πιο αυστηροί εμείς όσον αφορά τον ορισμό για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα άτομα στα οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα διευκρινίσουμε το θέμα της νομικής βάσης, θα το εξετάσουμε και στο Συμβούλιο, γιατί δεν αξίζει να συζητάμε στην οδηγία αυτή για συλλογικές συμβάσεις. Δεν παίζει ρόλο, γιατί αυτό το άτομα βρίσκεται ήδη στην επιχειρήση αυτή, είναι ήδη ε, υπάλληλος επιχειρήση αυτής. Άρα ισχύει ότι ισχύει. Και αυτό που θα έχουμε επιλέξει εκ των προ... επιλύσει εκ των προτέρων δεν χρειάζεται να το ξαναλύσουμε. Θα ισχύει αυτό που ισχύει στο κράτο μέλο ούτω ή άλλω. Αυτό θα είναι μια εξήγηση, μια λύση για τα πραγματικά προβλήματα, τα πραγματικά άτομα που έρχονται εδώ και δεν θα πρέπει κάθε φορά που μετακινούνται μέσα στην ίδια επιχείρηση από τη Γαλλία στην ε, Γερμανία ας πούμε να ξαναρχίζουν από το μηδέν σαν να μην είχαν ξαναμπεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγχος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχουν δικαίωμα τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ποιος μπαίνει στη χώρα τους και ποιος όχι. Αυτό το δικαίωμα των κρατομιλών θα πρέπει να διατηρηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους ελέγχους και είπαμε να μην ξεκινάμε κάθε φορά από το μηδέν. Και γι' αυτό θα πρέπει ο τρόπος με τον οποίο θα επιληθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα να έχει διακανονιστεί μεταξύ των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια της δέσμης για τη μετανάστευση. Και έτσι θα έχουμε μείωση των προβλημάτων, δεν θα έχουμε αυτή την ανάμιξη των διαφόρων αρχών, θα απλοστεύσουμε και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να σας πείσω να ακολουθήσετε αυτή την άγουσα. Η κυρία Γιασλόβιεσκα και ο κύριος Λάμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λαμβάνοντας αφορμή από όσα είπε η συνάδελφος, δεν καταλαβαίνω πώς θα διαχωρίσουμε στην πράξη την μετάθεση ενδοεπιχειρησιακός ε, σε σχέση με την ε, απόσπαση ας πούμε. Τέλος πάντων, εδώ τώρα να μην σας ε, καθυστερήσω, απλώς να αναφέρω ότι στις προτάσεις μας για την οδηγία αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρώπη θέλει να γίνει ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές, στο διεθνές προσκήνιο. Πρέπει λοιπόν να έχει μια αγορά εργασίας και υπεύθυνη αλλά και διαλεκτική ευέλικτη. Θα πρέπει λοιπόν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διασφαλίσουν καλές συνθήκες πρόσβασης των ειδικευμένων εργαζομένων, αυτών που έχουν υψηλά επαγγελματικά προσόντα. Η, μετά, μετάθεση, οι εσωτερικές αυτές αποσπάσεις, ας τις πούμε έτσι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να εξασφαλίσουμε την επαγγελματική κινητικότητα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Να μπορέσουν οι εργαζόμενοι δηλαδή να προσφέρουν τα προσόντα τους και σε άλλες χώρες. Υπάρχει έτσι καλή κυκλοφορία διαφορετικών γνώσεων, των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται και αυτό είναι σημαντικό τη σήμερα ημέρα. Το εργαλείο λοιπόν αυτό για την κινητικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να είναι και ζωντανό αλλά και να ε, επιτρέπει στους εργοδότες να αξιοποιήσουν τους εργαζομένους. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε στις τροπολογίες μας για την οδηγία αυτή στοιχεία που επιτρέπουν να αυξηθεί η ευελιξία. Για την ενδοεπιχειρησιακή κινητικότητα. Θέλουμε να υπάρχει μετάθεση εργαζομένων, δυνατότητα μετάθεσης, όχι μόνο για όσους έχουν εργασιακή σύμβαση, αλλά θέλουμε να προσφέρεται και μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας. Ο ορισμός για τους ειδικού, τους επαγγελματίες, να μετατραπεί ώστε να καλύπτονται και τα άτομα που ενδεχομένω η επιχείρηση να θεωρεί πλέον απαραίτητα σε μια άλλη χώρα. Το έθιξαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό εργαζόμενοι σε έναν όμιλο σε μια μεταβαλλόμενη αγορά να μην απασχολούνται αναδοδεκάμινο προτείνουμε για τους ε, εξειδικευμένους επαγγελματίες να μειωθεί το διάστημα αυτό σε έξι μήνες και σε τρεις για τους ασκούμενους. Επίσης θέλουμε να περιοριστεί η προθεσμία που προβλέπεται για την λήψη αποφάσεων. Είναι ιδιαίτερα μακρόχρονες οι αποφάσεις αυτές από 60 επιπλέον ημέρε θα θέλαμε να μειωθεί η προθεσμία αυτή σε 30 και από 80 σε 60. Αυτό τα διαστήματα είναι απολύτω επαρκή για να συγκεντρώσει κανεί τα απαραίτητα έγγραφα, τα χαρτιά του και να λάβει και την απόφασή του. Για τα θέματα τη κοινωνική ασφάλιση τώρα, το ανέφερε η κυρία Εσάγια τι γίνεται με τους μετατεθέμενους εργαζόμενους και την κοινωνική τους ασφάλιση. Στο άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο 2, στο εδάφιο C, δεν πρέπει να καλύπτουμε μόνο τις περιπτώσεις όπου μετατεθέμενοι εργαζόμενοι δίπτουν στο σύστημα το νομοθετικό μιας τρίτης χώρας για την κοινωνική τους ασφάλεια και τις εισφορές του. Δεν θέλουμε όμως να έχουμε περιπτώσεις εργαζομένων που τους καλύπτουν δύο ασφαλιστικά συστήματα και πληρώνουν δύο φορές τις εισφορές τους σε ένα τρίτο κράτος και σε ένα κράτο μέλος. Ε, εκεί που υπάρχει η ομοφωνία σε αυτήν την επιτροπή είναι ότι οι επιχειρήσεις που δρούν ανά την εφήριο καμιά φορά θέλουν να φέρουν το προσωπικό τους στις εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοητό αυτό αλλά αυτό που θέλουμε να φροντίσουμε είναι να αποφύγουμε τις καταχρήσεις. Πράγματα που γνωρίζω εγώ από τότε που ήμουν γενικό γραμματέα συνδικάτου. Να αποφύγουμε το μισθολογικό dumping, να αντικαταστούμε με φρέσκους Ινδούς ας πούμε το προσωπικό μιας επιχείρησης εδώ και επίσης αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι εξαιρούνται οι ασκούμενοι. Πρόκειται για ε, διοικητικό προσωπικό και θα αναφερθώ σε αυτό που είπε στην Αλφος Σουέτερ. Δεν ωφελεί τους εργαζόμενους μετά. Άμα θέλει να δει ποια είναι τα δικαιώματά του και δεν ξέρει ποια οδηγία, σε ποια οδηγία υπάγεται στην, για την ε, κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια σαφή νομική κατάσταση αν έχουμε κάτι καινούριο, μια νέα οδηγία για τους όρους εργασίας. Χρειαζόμαστε στην οδηγία αυτή και σαφή ορισμό ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι όροι που ισχύουν για αυτούς που έρχονται. Το θέμα της μετανάστευσης, αγαπητή κυρία Σρέτερ, δεν το συζητάω αυτή τη στιγμή. Εδώ διαφορόμαστε για το καθεστώς όσον αφορά την εργασία αυτών των ατόμων. Και έχω να πω ότι υπάρχει και ένα τομέα που δεν καλύπτεται από του ορισμού. Α πούμε, έρχεται κάποιο για έξι μήνε ε, ε, ε, από την Πολωνία σε μια εγκατάσταση μιας επιχείρησης και μετά πάει, τον στέλνουν μάλλον κάπου αλλού. Ε, δηλαδή τι θα ισχύει στην, στην ε, ε, περίπτωση αυτή. Θα ισχύει α, ο, θα ισχύουν οι όροι πληρωμής και λοιπά που θα έχει στην Πολωνία ή ε, εκείνοι που ισχύουν και για τους συνεργάτες του στην Γερμανία, Γαλλία όπου θα βρίσκεται. Αυτό πρέπει λοιπόν να το έχουμε απόλυτα ξεκάθαρο. Τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Καταλαβαίνω ότι οι κοινωνικοί εταίροι στην, στο τομέα των οικοδομών έχουν συμφωνήσει να μην ενταχθούν σε αυτή την οδηγία. Θα ήθελα όμως να αναφέρω πολύ προσεκτικά ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα πολιτικής, δηλαδή αν στο μέλλον έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες και ολόκληρη κλάδη δεν εντάσσονται στις ε, λόγω οδηγιες Εκεί θα έχουμε ένα νομοθετικό ευρωπαϊκό πρόβλημα και γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα στους κοινωνικούς εταίρους στο εθνικό επίπεδο, κατά πόσον υπάρχονται ή δεν υπάρχονται σε αυτή την οδηγία και να μην το εντάξουμε στην ε, κοινωτική νομοθεσία ότι υπάρχει μια εξαίρεση για ολόκληρο κλάδο οικονομικό. Ευχαριστώ. Πρώτος ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Η Επιτροπή θέλετε να διευκρινίσετε, μην επαναλάβατε τα προηγούμενα. Ίσως να διευκρινίσετε το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας περί μετάθεσης και τη διαφορά της σε σχέση με αυτήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγκεκριμένα για το σημείο που αναφέρατε. Να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη συντάσσουμε την πρόταση αυτή και κοιτάζουμε πολύ προσεκτικά το συσχετισμό μεταξύ του θέματος που συζητάτε με την οδηγία περιμετάθεσης εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών στον τομέα ICT δεν θα πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα από ότι οι Ευρωπαίοι υπήκοοι και εργαζόμενοι, όπως προβλέπονται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, αλλά και λιγότερα. Η κυρία Σάι έχει δίκιο. Όταν είπε ότι κάποιε φορέ οι εργαζόμενοι αυτοί de facto είναι και μετατιθέμενοι, άρα καλύπτονται από την οδηγία περί Ο κύριο Σέρκα είπε ότι μπορεί να είναι και ένα τη το ποσό που αφορά η κατηγορία αυτή. Εμεί όμω μπορούμε να πούμε ότι είναι 16.000 το χρόνο. Αυτό δείχνουν οι υπολογισμοί μας. Έχουμε άλλωστε και εργαζόμενους παρανόμως μάλλον που νομίμως διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οδηγία περί μετάθεσης προβλέπεται ότι εκείνο τους ή άλλους στο άρθρο 1 μπορούν να μετατίθενται από το ένα κάτω στο, ε, μέλος άλλο και για επικόους εργαζομένους μάλλον τρίτων χωρών στον τομέα ICT θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο με όσα προβλέπει η οδηγία για τις μεταθέσεις ενδοευρωπαϊκώ. Δηλαδή τι αυτηρές διτάξεις του άρθρου 1, τις βασικές διτάξεις του άρθρου 1 που θα πρέπει να καλύπτονται. Η οδηγία πάντως δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη εφόσον θέλουν να υπερβούν τα όρια αυτά να προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία στου ε, εργαζομένους τρίτων χωρών Αυτό όμω όχι βάσει τη οδηγία περί μετάθεσης, αλλά μόνο τη εθνική νομοθεσία. Αυτά έχω να πω για την ώρα. Το ευρωπαϊκό πρότυπο, νομίζω, μπορεί να μην είναι τέλειο, όπω ούτε και η οδηγία για τη μετάθεση των εργαζομένων, αλλά για την ώρα θα πρέπει να τα δεχτούμε. Η διαγραφή των παραπομπών στην οδηγία περί ε, μεταθέσεων δεν βελτιώνει την νομική ασφάλεια. Έχουμε δύο οδηγίε που αφορούν ακριβώ την ίδια κατάσταση. Για του σκοπού λοιπόν τη καλύτερη νομοθεσία και για την κάλυψη των αναγκών τη πραγματικότητα, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Η λύση που προτείνει η κυρία Σρέτερ είναι ελκυστική, αλλά δεν επιλύει το εγγενές πρόβλημα των μεταθέσεων και που προσπαθήσαμε με την οδηγία περιμετάθεση και τις διατάξεις της να το επιλύσουμε. Δηλαδή, μια εταιρεία ε, κατά πόσο έχει δικαίωμα να μεταθέτει του εργαζομένου τη ή όχι. Είναι το ερώτημα τη τα αυγό Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανεί απάντηση εδώ. Πάντω υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση και η Επιτροπή Προθυμία θα συνεργαστεί μαζί σα για να δούμε τη διασύνδεση της οδηγίας περί μετάθεσης εργαζομένων και του τι θα γίνει με τη μελλοντική πρόταση για την μετάθεση των εργαζομένων ICT από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η οδηγία αν δεν είναι τέλεια να την αναθεωρήσετε, έτσι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν θεωρείτε, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι τέλεια αυτή η οδηγία, αντί να μας λέτε ότι πρέπει να είμαστε πάντως να ζούμε ανάμεσά της μαζί της, τότε μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Να έχετε το λόγο. Ο κύριος Σέντελ έχει το λόγο πάλι. Ναι, ο εκπρόσωπος Κομισιόν είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε εργαζόμενοι που έρχονται βάσει των διατάξεων αυτών στην Ευρωπαϊκή να μην έχουν περισσότερο ή καλύτερα δικαιώματα. Μα πού ήταν ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν ε, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Δεν κατάλαβε αυτά που ηταν ο προσωπο τη κομισιον κατα τη διαρκεια τη συζητηση δεν καταλαβε αυτα που ειπαμε Δεν μα άκουσε. Μα δεν πρόκειται για το θέμα να έχουν περισσότερα δικαιώματα. Αγαπητοί κύριοι εκπρόσωποι τη Κομισιόν, πρόκειται για το θέμα τη αποφυγή των παραδάσεων και το θέμα του να μην έχουν οι άνθρωποι αυτοί λιγότερα, χειρότερα δικαιώματα. Μήπω θα μπορέσει η Κομισιόν να λάβει υπόψη και αυτή τη σκέψη. Πολύ καλά. Κύριε Σίγητα, συζητήσαμε για τόσα πολλά και διάφορα και παρακαλώ μην μακρηγορήσετε τόσο όπως πριν. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής δεν θα συζητήσω τα σημεία αυτά αλλά να μην είναι σίγουρο ότι είναι τόσο σαφές το πράγμα. Για το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ιδιαίτερα μπερδεμένο. Αυτό. Και αυτό σημαίνει σε εμά που θεωρητικά έχουμε μια κάποια μικρή γνώση. Εάν ε, το καταλαβαίνουμε έτσι εμείς, καταλαβαίνετε τι γίνεται απ' έξω που δεν το ξέρουν καθόλου. Σε ένα επίπεδο που αυτοί οι εργαζόμενοι είναι ο κριτικός λαβύρινθος με το μήνο, το μηνόταυρο, όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Το ίδιο, το διαφορετικό, αυτά είναι πολύ χειρότερα πάντως τώρα. Κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής, θεωρώ ότι είναι κάτι το απέσιο αφού μας εξηγήσατε από εδώ για το σημαντικό αυτής της δέσμης την ανάγκη που έχουμε γι' αυτό εντάξει δεν είναι σημαντικό είναι μόνο 18 εκατομμύρια στα οποία εφαρμόζεται αυτό. Τι γίνεται, μόνο για 18 εκατομμύρια ασχολείστε έτσι, τόσο ασχολείστε. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρότερο, σημαντικότερο. καταλαβαίνετε ότι πόσοι, αφορά το θέμα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιος είναι, ποιος μπορεί να μπει, κατά ποιες συνθήκες και να τελειώσουμε μια και έξω με το να δημιουργούμε την ίδια, τα ίδια προβλήματα με την προηγούμενη οδηγία για, για την εργασία. Έτσι θα πρέπει να μην έχουμε εκεί την μετάθεση των ίδιων προβλημάτων με την προηγούμενη. Και ορισμένα σχόλια ε, σίγουρα όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τη νομική βάση. Αν έχετε δίκιο κύριε Στρέτ, Στρέτερ, τότε η Λίσσα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να το εξετάσει έτσι. Ίσως θα πρέπει να δούμε τη νομική βάση από διαφορετικό πρίσμα. Δεν γίνεται αυτά τα θέματα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό όπως βλέπει το Συμβούλιο τα πράγματα δεν είναι το Συμβούλιο για την κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και η Επιτροπή και ο Επίτροπος Αρμός για την απασχόληση ότι είναι επικουρικός, βοηθητικός απέναντι στον άλλο και εμείς εδώ ότι είμαστε μόνο βοηθητικοί απέναντι σε άλλες επιτροπές. Έχουμε το θέμα της μετανάστευσης και το βασικό της πολιτικής μετανάστευσης και ενσωμάτωσης εδώ στην εργασία, στα εργατικά δικαιώματα, εργασιανικά δικαιώματα είναι κάτι το βασικό αποτελούν τη βάση της όλης ενσωμάτωσης και το αν είναι κανείς στο περιθώριο ή όχι. Από εκεί εξαρτάται και υπάρχουν ίσως άλλο προβλήματα με την διεύθυνση νομικής βάσης. Αλλάζουν οι όλες διαδικασίες οι νομοθετικές. Τέλος πάντων να το λύσουμε. Αλλά εδώ με τον κύριο εδώ της Επιτροπής εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι αυτισμός. Εδώ ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο και αυτό ε, ε, μας κάνει να, τους κάνει να γελάνε μαζί μας. Θα πρέπει να έχουμε κάτι το σαφές, το συγκεκριμένο, το διάφανο και όχι εδώ πολλά και διάφανο φορά και να καταλήγουν τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να λύσει περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν, εδώ η συγήτρια, η σωλιστική ομάδα, όλες αυτές είναι δυνατότητες και προς το παρόν φραστικά. Θα πρέπει να έχουμε, να έχουμε ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σαφώς να εκφράζονται οι σχέσεις ε, της οδηγίας αυτής με εκείνες της μετακίνησης των εργαζομένων. Κάτι ακόμα αυτά που είπαν στα αλήθεια Χίρς, ε, Σρέτερ, ε, Χροβιέσκ, ε, Χέντελ. Νομίζω ότι εκφράζουν πολύ καλά μια πραγματικότητα ότι όλοι έχουν αυτή τη διάθεση να πετύχουν μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των εταιριών, των επιχειρήσεων και στις ανάγκες των εργαζομένων και των κυρίων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί θα πρέπει να συγκλίνουμε στον δρόμο αυτό. Εδώ θα μπορούμε να πούμε, είδαμε ότι έχουμε αντιφατικές καταστάσεις. Αναφέρθηκε ότι αυτή η ομάδα εργαζόμενων, η εδώ ίσως ε, δεν ε, αποτελούν μία απειλή, ένα πρόβλημα για μια εκμετάλλευση εργασιακή. Ε, δεν έχουν να κάνουν, δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τους εργαζόμενους, τους εποχιακά εργαζόμενους που είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, εκείνοι αντιμετωπίζουν περισσότερο κίνδυνο, αλλά λιγότερος κίνδυνος για κοινωνικό ντάμπινγκ και στρεβλώσεις. Ε, εδώ θα πρέπει να δούμε αυτό το πλαίσιο με κάποια συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε τη διαφορά ανάμεσα αυτούς, γιατί αυτοί με ιδιαίτερε δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα μπορούν να προκαλέσουν τρομερή στρέβλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει βέβαια ένα κάποιο περιθώριο για τα κρατη αλλά ταυτόχρονα ε, βοηθάμε για ενέργειες δράση κατά της ασυμμετρίας, κατά της εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και παντού για όλους και για όλους όσους επωφελούνται από αυτό. Εδώ πιστεύω και Ακούστε να το σκεφτούμε γιατί σίγουρα έχει σχέση με οτιδήποτε εξετάσαμε μέχρι τώρα πολύ σωστά ακριβώς στις βόρειες χώρες ε, και στη δική σας ε, και στις υπόλοιπες ε, που έχουμε να κάνουμε αυτά για μεσολογικές εμβάσεις. θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όλα αυτά μέσω της οδηγίας των εργαζομένων, των μετακινούμενων γιατί το post-work εδώ αυτή η μετακίνηση αυτή καταστρέφει τη δυνατότητα των συλλογικών συμβάσεων, γιατί αυτό υπερισχύει απέναντι στα δικαιώματα αυτά μέσα των συλλογικών συμβάσεων. Γι' αυτό δεν νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι έχουμε αυτή τη διαφορετική, τόσο διαφορετική άποψη, αλλά θέλουμε, θέλουμε να γίνουν σεβαστές ε, οι εθνικές πρακτικές και σε μια ε, χώρα όπως τη δική σας που υπάρχουν τεράστιες απειλές είτε από ορισμούς είτε από κακούς ορισμούς αυτό το work και θα πρέπει να δούμε να μην μπει αυτός ο σπόρος της διχόνοιας ε, μέσω αυτών των συλλογικών συμβάσεων. Και τώρα κάτι τελευταίο. Να τονίσω κάτι. Η συγγήτρια, κύριε Κονσάρη, τι μου είπε έτσι έτσι έχουμε σε λίγο τις διακοπές. Αλλά σίγουρα θα εργαστεί, θα προσπαθήσει να διαβάσει τα πάντα, να δει ποια είναι τα θετικά και καταλαβαίνει ότι είναι αυτές απόψεις διάφορες ε, και να δούμε ποιες θα καταπέσουν, ποιες δεν είναι βάσιμες, αλλά ε, δεν θα υποστηρίξει μια σύγχυση, κάτι το άδικο και πολλά και διάφορα στα πλαίσια αυτών των τροπολογιών και που θα παλαμβάνει καταστάσεις όπως το παρελθόν. Θα πρέπει να νομοθετούμε καλύτερα και για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους, για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή μην ξεχάσει ότι έχει ζητήσει Τη έχει ζητηθεί μάλλον να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία αυτή σε τη διαστολή με την οδηγία περί μετάθεσης. Με το πιο ωραίο σας λοιπόν στυλό σημειώστε ότι θέλουμε μια απάντηση από τον Επίτροπο. Το δέχεστε? Χρειαζόμαστε διευκρίνηση για το σημείο αυτό. Λοιπόν, ναι, και το σημείωσα και θα το αναφέρω. Κι άλλο. ναι, αλλά ο εκπρόσωπο του άλλου επιτρόπου το σημείωσε. Διότι νομίζω ότι για τη μετάθεση εργαζομένων είναι η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης υπεύθυνη. Πρόεδρος, θέλουμε μια σαφή απάντηση για τη διάρθρωση μεταξύ των δύο οδηγιών. Και αυτό, εάν γίνεται σχεδόν με το κύριο του ίδιο του κυρίου Μπαρόζο Θέλουμε να έχει το κύρος, της, η απάντηση ολόκληρου του Κολεγίου των Επιτρόπων. Θέλουμε ο, ε, για να ικανοποιηθούμε όλοι μάλλον να δεσμεύονται από την απάντηση που θα μας απευθύνουν. Το σημειώσατε? Η Επιτροπή είναι αναγκαστικά κολέγιο. Non, non, mais le Parlement est aussi un Parlement et parfois nous connaissons des discussions. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε έντονε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται με στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό που ζούμε εδώ είναι ότι είμαστε ενωμένοι στην διαφορετικότητά μας. Λοιπόν, μπορούμε φαντάζομαι να έχουμε τη διευκρίνηση αυτή μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Euh, engagement. Alors... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Non C'est pas ça Si, c'est ça. Vous voulez reprendre la parole Θέλετε το λόγο πάλι. Α, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα το σημείωσα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να πάρετε την απάντηση ή τέλη Αυγούστου ή αρχή Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος. Ε, εντάξει, αρχέ Σεπτεμβρίου τα λέμε, δηλαδή 2 με 3 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, αλλά οπωσδήποτε μία απάντηση που θα δεσμεύει την πολιτική αρχή, όχι τι υπηρεσίε. Ωραία. Θα σα το δώσω και γραπτά. Γιατί αφού ζητάω εγώ τόσο υψηλή δέσμευση από την Κομισιόν, ε, νομίζω ότι καλύτερα να το στείλω αυτό γραπτά και στον αρμόδιο επίτροπο μάλιστα. και μετά θα πάω διακοπές. Λοιπόν, τούτον εχθένω θα εξετάσουμε τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες στις 19 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε από αυτόν στις 6 Οκτωβρίου. Και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσει και από αυτή τη έκθεση των... Ε, Νοέμβριο, όπως και για την έκθεση του κ. Κοφεράτη. Έχουμε το τελευταίο θέμα της σημερινής πρωίας. Στο σημείο 17 θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Φρανκ Έγγελ για τη διαδικασία αμοιβαίας εξολόγησης οδηγίας και τις υπηρεσίες. Έχει το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια που η διαδικασία μας για το θέμα αυτό ήταν στα αγγλικά, θα μιλήσω κι εγώ αγγλικά για τα δύο-τρία πράγματα που έχω να σας πω. Όπως συμβαίνει πάντα με γνωμοδοτήσεις, ε, πρόκειται για ένα σύντομα κείμενο. 1500 λέξεις ε, δικαιούμεθα. Δεν θα μας επιτρέπει κάτι τέτοιο να αναπτύξουμε τα θέματα. Αυτό που προσπάθησα να πω είναι μάλλον ε, επαναληπτικό σε σχέση με αυτό που έχει λεχθεί ήδη. Δεν είναι λοιπόν ε, επαναστατικό το κείμενο. Παρ' αυτά έχω μία σειρά τροπολογιών που μπορούν και να επιμηκύνουν το κείμενο τελικά. Το θέμα είναι ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς φαίνεται αποφάσισε να αναφερθεί πάρα πολύ στην διαδικασία της ε, αναθεώρησης ε, της αξιολόγησης. Και είναι λογικό. Πρόκειται για μια διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση. Καμιά άλλη ε, επιτροπή όμω δεν αποφάσισε να γνωμοδοτήσει και αυτό είναι σωστό μάλλον. Γιατί αν η δική μα επιτροπή αναφερόταν στην διαδικασία, θα είχαμε ξεπεράσει τα ωριά μας. Λοιπόν, θα πρέπει να αναφερθούμε στο περιεχόμενο αυτό για να σας εξηγήσω ότι ίσως δρούμε κατά κάποιο τρόπο παράλληλα με την Επιτροπή Επιστοσίας Ερμόδια. Για το κείμενο είδατε τι προτείνω. Σήμερα θα υποβάλω εγώ ίδιος δύο τροπολογίες που δεν ε, στρεβλώνω πολύ το κείμενο. Υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη με κάποια αριθμητικά στοιχεία με το τι, είναι, τι σημαίνει η υπηρεσία σε σχέση με το ΕΠ και την απασχόληση και σε σχέση με αυτό που καλύπτει σήμερα η οδηγία που είναι πολύ λιγότερα για να δείξουμε ότι πραγματικά υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης. Αυτά, κατά τα άλλα είμαι ανοιχτό ε, για οποιαδήποτε προσθήκη κλπ. κλπ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η κυρία Σαρμόδια Επιτροπή ασχολείται με τη διαδικασία και όχι με το περιεχόμενο. Πρόεδρος. Ωραία. Ακόμη και όταν συζητάμε το θέμα της λειτουργίας τη υπηρεσία της οδηγίας της υπηρεσίας, ε, υπάρχουν θέματα περιεχομένου. Κύριε Ντρονέν, πολύ σύντομα. Ίσως δεν διαφωνούμε και πάρα πολύ για το προτινόμενο κείμενο, για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Για το σημείο 3 όμως έχω ένα σχόλιο. Εκεί βλέπω να υπάρχει μια αντίφαση. Γιατί λέτε ότι ορισμένε υπηρεσίε έχουν αποκλειστεί από την οδηγία για τις υπηρεσίες λόγω της ειδικής του φύσης και ότι υπάρχει ε, δυνάμει ανάγκη για ε, κλαδική κοινοτική νομοθεσία. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτής της ιδέας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη ε, νομικής σαφήνειας και διευκρίνησης παν, μέσα στα πλαίσια της οδηγίας αυτής και γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια σημεία και να δώσουμε κάποιους συγκεκριμένους ε, ορισμούς, να υπάρχει δηλαδή νομική σαφήνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι η κλαδική κοινωτική νομοθεσία είναι χρήσιμη. Γιατί τι μιλάμε για φροντίδα παιδιών, δημοτικά σχολεία και τέτοια. θα υποβάλουμε κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ξέρω ότι το θέμα είναι αμφιλοκόμενο εδώ στο σώμα, αλλά ελπίζω ότι οι τροπολογίες μας θα είναι τόσο καλές που θα μπορέσουν πολλές συμφωνίες με αυτές σε ευχαριστώ. Κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έγγελ για την πολύ καλή πρόταση του. Ο συντάκτης της ε, νομοδότησης ξέρει ότι τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμη για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών θα πρέπει να ξεπεραστούν. Πρέπει ακόμα πολλά να γίνουν και ιδίως όσον αφορά στις δικές γιατί το 2 τρίτα του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχόλησης ε, προέρχονται από, την, ε, από τις υπηρεσίες, αλλά είναι μόνο το 20% του εμπορίου. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο από άδικη μεταχείριση. Γι' αυτό το 8% των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι δρούν και σε άλλες χώρες μέλη. Αυτό περιορίζει την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν όσον αφορά την αμοιβαία αξιολόγηση απαριθμεί τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχει παραδείγματο χάρη περιορισμός της συμμετοχή στα κεφάλαια και οι άλλες απαιτήσει που υπάρχουν. Η ανάγκη συνοχή στην εσωτερική αγορά για τι υπηρεσίε. Ε, παρεμποδίζει αυτή τη στιγμή την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς γιατί η, η οδηγία για τις περισσίες θα πρέπει να λάβει υπόψη και άλλες νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι ε, οι πρακτικές επιπτώσεις ε, της οδηγίας για τις αποσπάσεις και ποιες είναι οι επιπτώσεις για θέματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση και άλλα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης των διαμαχών. Εν τελευταία αναλύση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δράσουν. Οριζόντια νομοθεσία πλαίσιο δεν επαρκεί και οι διατάξεις ανακλάδο θα πρέπει επίσης να τροποποιηθούν. αν τα κράτη-μέλη και δύο χρόνια μετά την ε, ημερομηνία ε, εφαρμογή δεν ε, πληρούν τι υποχρεώσει, θα πρέπει να δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ και η Γκακούτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση όσον αφορά την πρώτη αξιολόγηση. Προσανατολίζεται περισσότερο στη διαδικασία όσον αφορά την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και εν μέρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Είναι η πρώτη εξολόγηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δούμε το 2011-2012 και ποια θα είναι η οικονομική αξιολόγηση της, της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς επίσης τον έλεγχο της απόδοσης όσον αφορά και τους καταναλωτές και τους προσφέροντες υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να είμαστε πλήρες αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις πτυχές. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να αναφερθούμε λιγάκι και στο περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πιο ευρύ χρήση, ε, να μην αναφερόμαστε δε στην συζήτησή μας μόνο για τις οδηγίες, στην οδηγία για τις υπηρεσίες, αλλά και άλλες οδηγίες που αφορούν την εσωτερική αγορά, όπως την μετάθεση κλπ. Να έχουμε δηλαδή την πλήρη εικόνα μπροστά μας θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες αλλά όχι ουσιαστικές. Γιατί σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την ε, γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ωραία. Η Κομισιόν δεν ζήτησε το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο. Θα ξαναδώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε για το δεύτερο αυτό γύρο. Περιγνώμη. Εγώ δεν διαφωνώ με κανένα από εκείνου που μίλησαν και του ευχαριστώ για τη συμβολή του. Θα ήθελα να πω στην κυρία Τουρουνέν ότι ναι. Συμφωνώ ότι ο όρος κεντρική κοινοτική νομοθεσία δεν είναι η ιδανικότερη διατύπωση και θα δεχθώ ευχαρίστως τροπολογίες που μπορούν να βελτιώσουν αυτή την ατέλεια. Ο λόγος για τους οποίους δεν αναφέρθηκα σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, οι κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή, οφείλεται στην... στο μέγεθος του κειμένου, στο μήκος του κειμένου και στον περιορισμό που έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί στο κείμενό μας όταν υποβάλλετε μια σχετική τροπολογία, οπωσδήποτε θα την υποστηρίξω. Και προς τον κύριο Κρότσμα και στην κυρία Κιόντς ε, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Μόνο ότι κατά γενικές σας, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τη γραφή που παρουσίασε. Και θα με βρούνε ευρέως συμφωνώ άμα υποβάλλουν αυτά που είπανε υπό μορφή τροπολογιών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που ολοκληρώσαμε έτσι τη συζήτηση για την παρουσίαση του σχεδίου σας γνωμοδότηση έχουμε μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών πολύ σύντομα μέχρι την επόμενη Τρίτη το μεσημέρι, 19 Ιουλίου δηλαδή για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ή μάλλον να συζητήσουμε στις 8 και να ψηφίσουμε στις 12 Σεπτεμβρίου. Τελειώσαμε τις εργασίες μας σήμερα το πρωί. Θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα.